Honorable Dear friends, can I ask all of you to take the seats? We would like to start our session. Πάρα πολύ καθίστε για να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Λοιπόν, καθίστε παρακαλώ, πρέπει να βάλετε και τα ακουστικά. Once again, dear friends, we are starting our session. Οι συνάδελφοι, θα αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Αγαπητοί φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά Επαναλαμβάνω με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω όλους τους παρευρισκομένους στην αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μάλιστα, κατά παράδοση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φιλοξενεί αυτές τις ημερίδες των ανοιχτών ημερών και ευελπιστώ ότι η ημερίδα αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μας βοηθήσει όλους όσοι συμμετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση, εκπροσώπους των κυβερνήσεων, των περιφερειών, των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, να προχωρήσουμε σε αυτές τις σκέψεις και τον προβληματισμό, γιατί προκλήσεις και ευκαιρίες έχουμε μπροστά μας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις που απαιτούν όχι μόνο μεγάλη σκέψη, αλλά και φιλόδοξες δράσεις. Θα εξετάσουμε λοιπόν κάποιες ε, απαντήσεις που θα δώσουμε μέσω των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές τις ε, ανοιχτές ημέρες γιατί μεσούς της κρίσης νομίζω ότι καλό είναι να βρούμε ένα χώρο που θα αφισβητήσουμε τις ε, προκαταλήψεις μας και θα διαρωτηθούμε κάποια θεμελιώδη ερωτήματα όχι μόνο για τις ε, προτεραιότητές μας αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το σωστό επίπεδο επίλυση των προβλημάτων είναι το τοπικό και, τοπικό και περιφερειακό παρόλο που οι ευκαιρίες ε, και οι προκλήσεις είναι πιο γενικές. Η αποτελεσματικότητα των δράσεων και των πολιτικών μας σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από την ανάμειξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και κάθε βαθμίδα διακυβέρνηση θα πρέπει να αναγνωρίσει ε, τις αδυναμίες ε, και τη, τα δυνατά της σημεία και να συνεργαστεί με τις υπόλοιπες βαθμίδες. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ για να συνεννοηθούμε και να συμφωνήσουμε για το κοινό μας έργο. Θα ήθελα να, να καλωσορίσω ολόθερμα τον Ζουζέ Μανώρη Μπαρόζο, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τον αντιπρόεδρο της Σουηδικής Κυβέρνησης που εκπροσωπεί την Σουηδική Προεδρία και είναι, Επίτροπος αρμόδια, είναι Υπουργός Αρμόδια για τις επιχειρήσεις. Επίσης θα ήθελα να καλωσορίσω και τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειών, τον Λουκ Βαντεμπράντε, καθώς και τον δόκτωρα Παύλ Σαμέτσκι που είναι ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα περιφερειακής πολιτικής και θα ήθελα να του δώσω το λόγο για σύντομες παρατηρήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, αγαπητοί φίλοι, ο Αντιπρόεδρος Μισελ Δελαμπάρ της Επιτροπής των Περιφερειών, κυρίες και κύριοι, Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι μεγάλη μου τιμή να σα συναντώ ξανά αυτή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τις Περιφερειές και τις Πόλεις ώστε να δούμε πάλι μαζί τον καθοριστικό ρόλο της συνοχής μεταξύ περιφερειακών και τοπικών εταίρων, την διαθεσμική συνεργασία, με σκοπό να οικοδομήσουμε την Ευρώπη στη βάση εταιρικών σχέσεων. Με το σεβασμό και την οικοδόμηση νέων δυνατοτήτων, ώστε όλοι να επενδύσουμε στην ε, ανάπτυξη των περιφερειών και των πόλων. Θα συνεχίσω στα Ολλανδικά. Η παρουσία σας και οι δεσμεύσεις σας σημαίνουν ότι η τωρινή εκδήλωση έχει μια ιδιαίτερη διάσταση. Βλέπουμε το βασικό εδώ ρόλο που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να αναλάβει, καταρτίζοντας την ε, πολιτική μας καθώς και η Επιτροπή, εκτιμώντας τον εδαφικό αντίκτυπο των αποφάσεών της. Επίσης, ε, χαιρετίζω την ε, νέα, τον νέο διορισμό του Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζου για δεύτερη φορά και μέχρι να συσταθεί πλήρως η νέα Επιτροπή θα πρέπει να σκεφτούμε και τη νέα εταιρική μας σχέση για το μέλλον. Και πάλι στα αγγλικά να συγχαρώ τον κύριο Μπαρόζο για το υπέροχο έργο του και θα μπορέσει να το συνεχίσει το εγχείρημα αυτό. Οι ευρωπαϊκές τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι άμεσα υπεύθυνε για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης που σωστά περιγράψατε αποτελεσματικές δράσεις για να βγει η Ευρώπη από την κρίση περιλαμβάνουν την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, την ανάπτυξη νέων πηγών για την βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, καθώς και την προώθηση της Ευρώπης των πολιτών. Βεβαίως, οι ανοιχτέ ημέρες, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι και μια πλατφόρμα για την ανοιχτή μας επικοινωνία, για διάλογο. Θα ήθελα εδώ να αποτίσω φόρο τιμής στον ε, κύριο Σαμίτσι, για έβδομη φορά για την ε, υπέροχη συνεργασία που είχαμε με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειών. Επιτρέψτε μου να πω εκ μέρου τη Επιτροπή των Περιφερειών πόσο ικανοποιημένοι είμαστε με τα θετικά αποτελέσματα του Ιρλανδικού δημοψηφίσματο. Δεν μπορώ παρά να επαναλάβω τα λόγια του κυρίου Μπαρόζο. Σε ευχαριστούμε Ιρλανδία. Thank you Ireland. Οι ειδήσει είναι πολύ καλέ για όλου μα και για την εδαφική συνοχή. Η νέα συνθήκη θα θέσει τα θεμέλια για μια πιο δυναμική, δημοκρατική και διαφανή ένωση. Θα είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του μέλλοντος και για τις χώρες μας και για τον κόσμο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ανοιχτές ημέρες, να αναφέρω μόνον ορισμένα από τα βασικά σημεία τα οποία θα λάβουν χώρα τις επόμενες ημέρες. Τα κράτη-μέλη και η Ευρώπη πρέπει να βασίζονται στους περιφερειακούς και τοπικούς εταίρους και για την περιφερειακή, απόκριση στην οικονομική κρίση χρειαζόμαστε τις τοπικές απαντήσεις για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και την εδαφική συνεργασία για να στηρίξουμε γενικότερα τη συνεργασία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καλύτερη ποιότητα ζωής. Πρώτον, οι περιφερειακές αποκρίσεις στην οικονομική κρίση είναι ε, μέρος ενός σαφούς μηνύματος. Ο αντίκτυπος της κρίσης μπορεί να ποικίλει από τη μια περιφέρεια στην άλλη. Οι λύσεις όμως θα εξαρτηθούν από την περιφερειακή δράση. Οι λύσει θα εξαρτηθούν από την περιφερειακή δράση, επαναλαμβάνω. Οι περισσότερε προκλήσει που σήμερα απασχολούν τι τοπικέ και περιφερειακέ κυβερνήσει δείχνουν ότι υπάρχει εδαφική διάσταση, ισχυρή εδαφική διάσταση για τι περισσότερε περιφέρειες και πόλει. Η κρίση θα αυξήσει την έκθεση στι παγκόσμιε αγορέ οι αποτυχίε των επιχειρήσεων, οι απώλειε θέσεων εργασιών, η πίεση στου προπολογισμού των κρατών και η ανάγκη να γίνουμε πιο καινοτόμοι είναι θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή των Περιφερειών αύριο θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα των διαβουλεύσεών τη, που ξεκίνει με σκοπό την, το νέο σχεδιασμό της στρατηγικής της Λισαβόνας για το 2010, ώστε 80 εταίροι και συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία και αυτοί να δώσουν τη συνεισφορά τους σε αυτή την ε, σχεδιασμό το νέο σχέδιο περιφερειακό και τοπικό εγχείρημα της Ευρώπης έχει σκοπό να προωθήσει και το επιχειρήν σε ευρωπαϊκό και τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Εδώ στόχος του Συμβουλίου είναι να δείξει και ένα βαθμό ευελιξίας ως προς την συγχρηματοδότηση και για να αντιμετωπιστούν έκτακτες συνθήκες όπως αυτές τις οποίες συχνά αντιμετωπίζουμε. Έπειτα, οι ανοιχτέ αυτέ οι θα αποδείξουν ότι οι περιφέρειε, οι επαρχίε και οι πόλει τη Ευρώπη είναι ενεργοί εταίροι στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Πολλέ από αυτέ ήδη έχουν πρασινότερε τοπικέ οικονομίε. Χρειάζονται όμω και κρατικέ διευκολύνσει και στηρίξη από τον προπολογισμό. Οι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ πρέπει να γνωριστούν και να ανταλλάξουν βέλτιστε πρακτικέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την πρόληψη, την προσαρμογή, την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και τι βιώσιμε μεταφορέ. Γι' αυτό οι περιφέρειε και πόλει τη Ευρώπη θα είναι παρούσε στην Σύνοδο για τι Κλιματικέ Αλλαγέ στην Κοπενχάγη του ΟΗΕ. Επίση θα συνεχίσουν τι κλιματικέ αλλαγέ να θεωρούν ως μία πρώτη προτεραιότητα και πέραν τη Συνόδου της Κοπεχάγης. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε προσκαλέσει τον μελλοντικό πρόεδρο της Συνόδου την επόμενη Τετάρτη ώστε να διερευνήσουμε τις δυνατότητες ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Έπειτα, η συνεργασία μεταξύ των περιφερειών, των ε, διαφόρων εδαφικών τμήματων τη Ευρώπη. Είναι ένα πραγματικό παράδειγμα ότι η, Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Η διασυνοριακή συνεργασία. Η στρατηγική για τη Βαλτική θάλασσα και άλλες πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες, όλες έχουν τέτοια εμβέλεια που ε, μπορούν να ακολουθηθούν και από άλλα παραδείγματα στη Βόρεια Θάλασσα και αλλού. Οι συζητήσει αυτέ λοιπόν έχουν δώσει αφορμή για πολλέ εκδηλώσει, οι οποίε θα εκτεληθούν και τι ερχόμενε ημέρε και θα αποδείξουν το πραγματικό ενδιαφέρον των τοπικών αρχών. Τέλο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, το μελλοντικέ προτεραιότητε και ο προπολογισμό τη Ένωση θα εντατικοποιηθούν σύντομα. Η πολιτική δαφική συνοχή θα συνεχίσει να είναι ανοιχτή σε όλε τι περιφέρειες. Ανοιχτή σε όλε τι περιφέρειες, επαναλαμβάνω θα, δεν θα υπάρχουν αυτοί που κερδίζουν ή χάνουν ω προ την οικονομία. Θα πρέπει όμω να αντιμετωπίσουμε από την άλλη και τις, ε, τον αντίκτυπο τη παγκοσμιοποίηση, τη δημογραφική πίεση και τη οικονομική κρίση. Η αυριανή πολιτική συνοχή θα πρέπει να ενισχύσει τι δυνατότητε για την βιώσιμη ανάπτυξη όλων των περιφερειών, βελτιώνοντα τι δυνατότητε καινοτομία, το επιχειρήν, την βιωσιμότητα, την απασχόληση και την προσβασιμότητα. Επιπλέον, η διδαφική συνοχή θα πρέπει να ε, αντιμετωπίζεται ως μια νέα δυνατότητα ελευθερίας για τους πολίτες μας. Ελευθερία να επιλέξουν πού θα ζήσουν τη ζωή τους και πού θα εργαστούν άσχετα από γεωγραφικές ε, αναπηρίες ή περιορισμούς. Πρέπει να γίνει ένα εργαλείο που θα μετατρέψει την εδαφική ποικιλότητα σε περιφερειακή δύναμη. Η Ευρώπη δεν μπορεί να γινει ενα εργαλειο που θα μετατρεψει την ανταφική ποικιλοτητα σε χωρίς τις περιφερειές και τις πόλεις της, όποιο και αν είναι το ζήτημα που την απασχολεί. Κανεί δεν μπορεί να χτίσει ένα σπίτι ξεκινώντα από τη στέγη. Οι περιφέρειε και οι πόλεις της Ευρώπης θα πρέπει να, να αντιμετωπίζονται ω τα στέρεα θεμέλια που μπορούμε να χτίσουμε την ένωσή μα βασισμένη σε μια σχέση εταιρική, πραγματικά εταιρική. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Like Σας ευχαριστώ τώρα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον δόκτωρα Πάβελ Σαμέτσκι, τον αρμόδιο επίτροπο για θέματα περιφερειακής πολιτικής. Κυρία Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, μέλη της Επιτροπής Περιφερειών, εκπρόσωποι της ε, τοπική και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, σας καλωσορίζω θερμά στην έβδομη αυτή διοργάνωση των Open Days και οι χιλιάδε καλεσμένοι μα από τους ακαδημαϊκούς του επιχειρηματικού κύκλους, τα μέσα μαζική ενημέρωση ε, τη Ευρώπη και του κόσμου, εκπροσώπους των ΗΠΑ, τη Ρωσία, της Κίνας, της Βραζιλίας, της Ουκρανίας. Ε, η συμμετοχή αυτών των αξιότιμων προσκεκλημένων ε, καθιστούν αυτή την οργάνωση το μείζον γεγονό για τις περιφέρειες. Η περιφερειακή πολιτική χορηγεί πολλά κονδύλια και ενισχύει τι επενδύσεις και επιτρέπει στου ανθρώπου από τι διάφορε περιοχέ τη Ευρώπη να αναζητήσουν του καλύτερου τρόπου για την ανάπτυξη των περιφερειών του. Από τι περσινέ Open Days ε, πολλά έχουν ε, συμβεί. Αντιμετωπίσαμε την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση με την οποία ε, απαντήσαμε προτείνοντα το Ευρωπαϊκό Σχέδιο οικονομική ανάκαμψη, καθώ και διάφορα άλλα εθνικά και περιφερειακά μέτρα και προσπαθούμε να εστιάσουμε τι τωρινέ αυτέ Open Days στις ε, παγκόσμιες προκλήσεις και τις ευρωπαϊκές απαντήσεις αυτές. Θέλουμε έτσι να προβούμε σε μια ανταλλαγή απόψεων και να δεχθούμε καλύτερα από τις εμπειρίες μας για να δούμε πώς θα περάσουμε αυτή τη δοκιμασία οι περιφέρειες, πώς θα μετατρέψουμε την πρόκληση σε ευκαιρία. Και έχουμε ως βασικά θέματα την καινοτομία, τις κλιματικές αλλαγές, την εδαφική συνεργασία και το μέλλον της πολιτικής ε, συνοχής. Καταρχήν, το θέμα της καινοτομία. Η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση έχει δύο από τις τρεις πιο καινοτόμες χώρες του κόσμου στους κόλπους της. 17 όμως ε, χώρες μέλη δυστυχώς βρίσκονται κάτω από τον κοινοτικό μέσο όρο. Παρόμοιες ανισότητες ε, και χάσματα υπάρχουν και μεταξύ των περιφερειών. Οι μισές από τις ευρωπαϊκές περιφέρειες ε, αντιμετωπίζουν τεράστιο χάσμα σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις τους στις καινοτομίες. Γι' αυτό αυτό το χάσμα θα πρέπει να γεφυρωθεί. Αυτό είναι πρόκληση της κοινωνικής συνοχής, γιατί μέχρι το 2013 θα ε, επενδύσουμε γύρω στα 90 δισεκατομμύρια, δηλαδή λιγότερο από το 1 τέταρτο της ε, περιφερειακής πολιτικής σε θέματα καινοτομίας. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια για να επαναφέρουμε την αηφόρο ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερη πρόκληση, κλιματικές αλλαγές. Οι ευρωπαϊκές δεσμεύσεις στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών ζητά από τι ε, περιφέρειε να αναμορφώσουν τι οικονομίες του ιδιαίτερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρε. Με τι Open Days αυτέ, ε, θα δούμε ποιε είναι οι βέλτιστε πρακτικέ και ποιε είναι οι καλύτερε τοπικέ και περιφερειακές προσεγγίσει για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, προκειμένου να δούμε πω η περιφερειακή πολιτική θα συμβάλλει αποτελεσματικά σε μια αηφόρο οικονομική ανάπτυξη. Ένα άλλο μείζον θέμα των φετινών Open Days είναι η εδαφική συνεργασία η περιφερειακή συνεργασία. Φέτο ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτησε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την περιοχή της Βαλτική. Αυτό το νέο κεφάλαιο δίνει έναν ε, νέο τρόπο συνεργασίας και ε, μπορούμε αυτή την ε, μακροπεριφερειακή προσέγγιση να τη μεταγγίσουμε και σε άλλε πολιτικέ τη Ένωση. Θα έχουμε συζητήσει με στρατηγικούς μας εταίρους για να δούμε πώ θα συνεργαστούμε με το πιο αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου αυτή η συνεργασία τη Βαλτική να γίνει υπόδειγμα για συνεργασία σε άλλες περιοχές όπως ε, του Δούναβη. Το τελευταίο θέμα των Open Days είναι το μέλλον τη πολιτική συνοχή. Μάλιστα πρόσφατα ολοκληρώσαμε κάποια αξιολόγηση των προγραμμάτων 2000-2006 που καταλήγουν στην αδιαφυσβήτητη προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά επιστούν την ανάγκη αλλαγής, προκειμένου να προσανατολιστούμε περισσότερο προς τα αποτελέσματα και να πλουστεύσουμε καλύτερα τις διαδικασίες. Η προκάτοχός μου, Ντανούτα Χιμπνέρα, γεννήσε σημαντικές συζητήσεις για το θέμα αυτό, που είναι ιδιαίτερα προσφυλές και σε μένα και με βάση τις συζητήσεις αυτές θα εκπονήσω ένα έργο ανατολισμό για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής. Και στα πολυάριθμα σεμινάρια που θα γίνουν εδώ θα λάβουμε και εμείς πολλές προτάσεις και ιδέες. Θέλουμε αυτή η οργάνωση των Open Days να γίνει ένα είδος γνωστικής διαδικασίας γιατί θα έχουμε πάνω από 60 κορυφαίους ακαδημαϊκούς από πολλές ε, περιοχές του κόσμου που θα μας ε, διαφωτίσουν για τα διάφορα θέματα. Επίσης, στο δρόμο αρσιμέντ έχουμε το περίπτερο της, των Open Days. Εκεί θα γίνουν πολλές εκθέσεις και happenings. Σας προσκαλώ να το παρακολουθήσετε στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Τέλος, ήθελα να ευχαριστήσω θερμά σε όλους όσους κύριους συνέβαλαν στην προετοιμασία αυτών των ανοιχτών ημερών του 2009. Η οργάνωση αυτή κατέστηκε χάρη στην ανοιχτή ε, και επικοδομητική συνεργασία μεταξύ των εταίρων τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακή Πολιτική τη Επιτροπής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, καθώ και τι ε, περιφέρειες και πόλεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα γραφεία του στην Ευρώπη. Σας εύχομαι καλή τύχη για την εβδομάδα αυτή σε όλους όσοι συμμετέχουν στα σεμινάρια και τα εργαστήρια και ελπίζω να εκμεταλλευτείτε τη γνώση αυτή, τις ιδέες και τις εμπειρίες που θα ανταλλάξετε όλες αυτές τις μέρες επεξεργαστείτε τες, μεταβιβάσετε στην πατρίδα σας και διαβιβάστε και μεταδώσετε τες περαιτέρω. Thank Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ε, τελειώσαμε τις ε, εισαγωγικές ομιλίες για το καλωσόρισμα στα εγγένεια των Open Days και τώρα θα δώσω τον ε, λόγο στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Μανουέλ Μπαρόζο, για τη δική του ομιλία. Monsieur Περιφερειών, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής ε, για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κυρία Αντιπρόεδρε της Σουηδίας που αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί το Συμβούλιο, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι. Είμαι πολύ ευτυχής που μπορώ να λάβω μέρος ε, στην έναρξη των Open Days. Ε, είμαι ένας θαμώνας ε, αυτών των εκδηλώσεων που είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικές και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή των Περιφερειών και επίσης και τον Επίτροπο της Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη Γενική Ανάπτυξη και την Επιτροπή ανάπτυξης. Έρχομαι από το Pittsburgh ε, και από την συνέντευξη και από την διάσκεψη της ε, Νέας Υόρκης. Ε, πρόκειται για δύο πολύ σημαντικά παγκόσμιες συναντήσεις, για δύο πολύ σημαντικά θέματα, δηλαδή για την καταπολέμηση της ανεργίας και για το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Και βεβαίως ε, αυτά είναι τα θέματα τα οποία διαλέξατε κι εσείς ε, για τις ε, Open Days, δηλαδή για την κρίση της παγκοσμιοποίησης και για τις περιφερειακές απαντήσεις. Θα πρέπει να δώσουμε νέες απαντήσεις γιατί ο κόσμος ο οποίος θα βγει από την κρίση δεν θα είναι πια ο ίδιος, θα έχει ανάγκη από νέους κανόνες και ακριβώς αυτό είναι το πολιτικό ζητούμενο. Και βεβαίως ε, το, ο κύριος στόχος μας είναι να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την ε, κρίση. Βεβαίως υπάρχουν όλα αυτά τα προγράμματα ανάπτυξης. Ε, θα πρέπει να υπάρξει μια τεράστια προσπάθεια στα πλαίσια του προπολογισμού. Θα πρέπει να πούμε ότι ένα πέντε ένα 5% του ΑΕΠ αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται και θα πρέπει να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ποσοστό σε πολλά ε, επίπεδα ε, για την ε, καταπολέμηση της ανεργίας θα πρέπει επίσης να υπάρξει μια βελτίωση των υποδομών και θα πρέπει να υπάρξει μια ανάκαμψη. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει μια καινούργια δυναμική παγκόσμιου χαρακτήρα στα πλαίσια του 20 για να μπορέσουμε να λάβουμε μέτρα που θα καταπολεμήσουν την κρίση και που θα έχουν βεβαίως και οικονομικό ε, χαρακτήρα. Ε, και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση και στο Facebook προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε αυτή την δυναμική των διαβουλεύσεων και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας έλεγχος και μια πολύ σημαντική συνεισφορά για την παγκόσμια οικονομία γιατί θα έλεγα ότι ενστικτοδός και φυσικό τον τρόπο είμαστε υπέρ μιας παγκόσμιας διαχείρισης και διακυβέρνησης. Εκτός από τα έκτακτα μέτρα θα πρέπει να υπάρξει μια ε, ένα προγραμματισμό ο οποίο θα είναι μακροπρόθεσμο και θέλουμε αυτή τη στιγμή να υπάρξει μια, ένας νέος προγραμματισμός ο οποίο θα έχει ηθικό χαρακτήρα και θα είναι πιο αξιόπιστο. Οι πραγματικέ οικονομίε έχουν ανάγκη. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να μπορεί να, προ, να υποβάλει προτάσεις όπως έγινε στο Πίτσπουργκ. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό σύστημα οικονομική εποπτεία και οι προτάσεις νομικού, νομοθετικού περιεχομένου αυτή τη στιγμή θα προταθούν στα πλαίσια του Συμβουλίου. Είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι μπορέσαμε να υποβάλουμε προτάσεις ε, νομοθετικού περιεχομένου στο Πίτσμπουργκ. Και βεβαίω δεν φτάσαμε στο τέλο του τούνελ. Ξέρουμε ότι η οικονομική κρίση ε, δεν έχει τελειώσει και υπάρχουν πολλέ ε, κοινωνικέ εντάσει, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να σταματήσει η ελεύθερη πτώση, έχει σταματήσει αυτή η ελεύθερη πτώση της οικονομίας, υπάρχει μια μικρή ανάπτυξη, μια μικρή ανάκαμψη της οικονομίας και αυτό παρατηρείται στο δεύτερο εξάμεινο του 2009. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα ε, μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε την ανάπτυξη τη στιγμή που αυτή τη στιγμή αυξάνεται η ανεργία. Και κατά την άποψή μας δεν υπάρχει μια πραγματική ανάκαμψη τη στιγμή που αυξάνεται η ανεργία. Η ανεργία, κατά πολέμηση ανεργίας αποτελεί το κύριο μέλημά μου γιατί πλήττει τους πιο ευάλωτους, τους ανειδίκευτους, τους νέους ε, και τις ευαίσθητες κατηγορίες του πληθυσμού, δημιουργεί τον κοινωνικό αποκλεισμό, ε, την ανέχεια, την παινία. επίσης ε, θέτει σε κίνδυνο τον, την κατανάλωση, θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρξει μια γενική κινητοποίηση για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την ανεργία στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ακολουθεί το δρόμο της. Υπάρχει ένα πρόγραμμα ανάκαμψης, ανάπτυξης και βεβαίως υπάρχουν ε, και πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν διατεθεί θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους νέους ε, οι οποίοι είναι ανειδίκευτοι αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να υπάρξουν προτάσεις για το μέλλον και χρειάζεται μία ε, συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων στα πλαίσια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κοινωνικών εταίρων, των χωρών μελών σχετικά με την κατάρτιση, με την ανάπτυξη. Η οικονομία της γνώσης θα πρέπει να αποτελέσει μία προτεραιότητα και επίσης έχουμε απλοποιήσει τη διαδικασία σε σχέση με τα διαφορετικά ταμεία και σε σχέση με την ροή των κονδυλίων θέλουμε να βοηθήσουμε αυτούς που είναι άνεργοι αυτή τη στιγμή για να έχουν ξανά πρόσβαση στο χώρο εργασίας. Επίσης υποβάλαμε μία πρόταση σχετικά με τις συνθήκες της χρηματοδότησης που ε, θα μπορέσει να, να αντιμετωπίσει την κρίση. Επίσης θα πρέπει το Συμβούλιο να δεχθεί αυτές τις προτάσεις και είναι προφανές ότι σε μια τέτοια κατάσταση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε θα χρειαστούμε περισσότερη ευελιξία σχετικά με την χρήση των κονδυλίων των διαφορετικών ταμείων. Και αυτό οι περιφέρειες το γνωρίζουν πολύ καλά. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι αυτή τη στιγμή αποφασίσαμε να υπάρξουν 50 εκατομμύρια ευρώ, μια ε, ροή ε, κονδυλίων που θα βοηθήσουν τους άνεργους να ιδρύσουν τις δικές τους επιχειρήσεις και ακριβώς αυτό θα μπορέσει να βοηθήσει την ανάπτυξη. Ε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη της ε, ε Επιτροπής των Περιφερειών και αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα απλώς να σας πω ότι στα τέλη της περασμένης εβδομάδας πήραμε πολύ καλές ειδήσει από την Ιρλανδία. Η Ιρλανδία είπε ναι στην Ευρώπη, ψήφισε ναι για την Ευρώπη. Νομίζω ότι η απόφαση αυτή τη φορά του Ιρλανδικού λαού ήταν μια αναγνώριση ότι η Ιρλανδία έχει επωφεληθεί από την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Ο λαό τη Ιρλανδία αναγνώρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι, πράγματι ήταν ένα σημαντικό παράγοντα για την αντιμετώπιση της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Βέβαια, λόγος για την κρίση πρέπει να γίνει. Όμως κάποτε αυτή η κρίση θα είναι μια δυσάρεστη ανάμνηση και όσο πιο γρήγορα έρθει αυτή η μέρα τόσο το καλύτερο. Εν τω μεταξύ πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την ανάκαμψη. Πρέπει να συνεχίσουμε να ετοιμαζόμαστε για το μέλλον. Οι πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές που παρουσίασα τις επόμενες, πριν από λίγες μέρες για την ερχόμενη θητεία της Επιτροπής και λίγες μέρες μετά την εκλογή μου θα στηριχθούν βεβαίως από το Ευρωκοινοβούλιο και καθορίζουν μια συνολική θεώρηση για την Ευρώπη με έναν χρονικό ορίζοντα ως το 2020, ώστε να μετατραπεί η Ευρώπη σε μια πράσινη οικονομία μια οικονομία της γνώσης, μια βιώσιμη οικονομία που να επικεντρώνεται στην κοινοτομία. Εάν υλοποιήσουμε αυτή την πολιτική θεώρηση, αυτό σημαίνει ότι μετά το 2010 θα πρέπει να έχουμε εντωμεταξύ μεταρρυθμίσει και τη στρατηγική της Λισαβόνας. Η Επιτροπή των Περιφερειών πρόσφατα συνέταξε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση για το μέλλον αυτής της στρατηγικής. Αυτό που θα πείτε εσείς και η δική σας γνώμη για μας είναι πολύ σημαντικό. Δεν είσαστε απλώ οι διαχειριστέ των ε, διευθυντικών ταμείων. Έχετε κοινή ευθύνη για τι πολιτικέ που καλύπτονται από τι κοινέ μα στρατηγικέ για την ε, ανάπτυξη και την έρευνα, την καινοτομία, το επιχειρηματικό περιβάλλον, την εκπαίδευση, την διαβίωμάθηση, τι τις μεταφορές, την ενεργειακή αποδοτικότητα. Πραγματικά χρειαζόμαστε την δέσμευση και τη συμμετοχή των περιφερειακών αρχών ε, και των τοπικών αρχών και των επαρχιών. Χρειαζόμαστε τις δικές σας γνώσεις και τις θετικές σας εμπειρίες. Γνωρίζουμε καλά ότι η επιτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας για το διάστημα μετά το 2010 σε όλη την Ευρώπη θα εξαρτηθεί από εσά. Αυτή η στρατηγική θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναδυθούμε από την κρίση και να αναλάβουμε πρωταρχικό ρόλο στο να κάνουμε την, το όραμά μας αυτό πραγματικότητα. ώστε να υπάρχει μια οικονομία της αγοράς σφαιρική, η οποία να δίνει τη δυνατότητα συμμετοχή σε όλους, να είναι ενδιαφέρουσα για τους επενδυτές και να ε, γύρει το πνεύμα του επιχειρήν. Μια κοινωνία ανοιχτή που να προωθεί την καινοτομία, να δίνει απασχόληση στους πολίτες, να δίνει ευκαιρίες για έρευνα και τεχνολογία. Να επενδύει στην κοινωνική συνοχή. Να δίνει πραγματικά δυνατότητες για διαβίου μάθηση και να επιτρέπει την πιο οικολογική αντιμετώπιση πολλών οικονομικών τομέων. Αυτή η αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο εάν συμπληρωθούν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι ότι πρέπει όλοι να συνεργαστούμε. Πρόσφατα Μίλησα για την εταιρική σχέση που χρειαζόμαστε για την πρόοδο. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε από κοινού τι προκλήσει που έχουμε, όλοι οι συμμετέχοντε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά όργανα, οι τοπικέ αρχέ, οι περιφερειακέ αρχέ, οι κυβερνήσει, οι κοινωνικοί εταίροι, οι πολίτε, πρέπει όλοι να κινηθούμε μαζί στην ίδια κατεύθυνση και να αγωνιστούμε, όπω είπε ο πρόεδρο Βάντεμπραντε, και το γνωρίζει πολύ καλά, δεν το λέω σήμερα μόνο και μόνο επειδή μιλώ μπροστά σα στην Επιτροπή των Περιφερειών. Είναι πραγματική μου πεποίθηση ότι μόνον συνεργαζόμενοι σε εταιρική σχέση σε όλα τα επίπεδα λήψη αποφάσεων μπορούμε να κάνουμε την Ευρώπη να ζήσει αυτό το όραμα που έχουμε σχεδιάσει. Και ορίζοντα πενταετία που έχουμε μπροστά μα θα αντιμετωπιστεί από κοινού με το Ευρωκοινοβούλιο. Χωρί αυτή την εταιρική σχέση και τη συνεργασία δεν θα είχαμε πετύχει ούτε τώρα ούτε στην Ιρλανδία. Και να σα πω ότι ήμουν, ήμουν και εγώ εκεί, στο Λίμερικ. Και δεν ήταν ένα θέμα του κράτους μόνο, δεν ήταν ένα θέμα των κομμάτων το δημοψήφισμα αυτό. Είχαν συμμετοχή όλα τα επίπεδα της κοινωνίας των πολιτών. Γι' αυτό να δώσουμε μεγάλη πλειοψηφία των Ιρλανδών ψήφισαν υπέρ με τόση σαφήνεια για την Ευρώπη. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη προϋπόθεση να επενδύσουμε σε νέες πηγές βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε με μερικές από τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες όπως η Ινδία, η Κίνα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα ίδια παλιά εργαλεία που είχαμε τώρα στη φαρέτρα μας. Πρέπει να αναζητήσουμε νέες ε, λύσεις. Πράσινη οικολογία, νέα τεχνολογικά μοντέλα, μελλοντικά δίκτυα, υποδομές, τεχνολογία. Και εδώ θα δούμε τη δεύτερη μεγάλη πρόκληση που σα ανέφερα προηγουμένω τι κλιματικέ αλλαγέ. Εδώ έχουμε ηγετικό ρόλο στο διεθνέ προσκήνιο, γιατί είμαστε αποφασισμένοι, αποφασισμένοι να προχωρήσουμε. Έχουμε ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο που είναι παράδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο και εμείς οι Ευρωπαίοι δώσαμε το ρυθμό στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Είναι λοιπόν καθοριστική σημασία οι εταίροι μα να μας ακολουθούν, οι Ηνωμένε η Ιαπωνία, επιταχύνουν την κίνησή τους προς μια κοινωνία και οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα. Πρέπει να επιμείνουμε λοιπόν σε αυτό, αλλά θα πρέπει να είμαστε και Ενεργεί στι διαπραγματεύσει που γίνονται ω τώρα. Ε, Κυρίε και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση στι περιφέρειε, τι επαρχίε και τι πόλει τη πρέπει να επενδύσει ώστε να διατηρήσει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και να παραμείνει και ανταγωνιστική στο διεθνέ προσκήνιο. Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι εχθρό τη επικουρικότητα. Στην πραγματικότητα, το ακριβώ αντίθετο αληθεύει οι περιφέρειες είναι ακριβώς το σημείο που μπορεί να αποκτηθεί γνώση, να αναπτυχθεί η οικονομική αντιδραστηριότητα, να αναπτυχθεί απασχόληση, κοινωνική συνοχή και τα καινοτόμα συστήματα. Ο στόχος της πολιτική συνοχής είναι ακριβώς να καλλιεργήσει την ευρωπαϊκή ε, αλληλεγγύη και να ενθαρρύνει τις περιφέρειες να αντιμετωπίσουν τι διάφορε προκλήσει που υπάρχουν. Γι' αυτό λοιπόν Νομίζω ότι βρισκόμαστε στην αρχή ενό νέου κύκλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ερχόμενη πενταετία. Πιστεύω πολύ στο μέλλον τη πολιτική συνοχή και τη περιφερειακή πολιτική. Τα στοιχεία αυτά είναι αποφασιστική σημασία για το πώ θα καθορίσουμε τη νέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. I would like to thank President... Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζωζε Μανώλη Μπαρόζο, όχι μόνο για την παρουσία του σήμερα εδώ, αλλά για το γεγονός ότι τελευταία πενταετία ήταν συστηματικά μαζί μας ε, στις εβδομάδες ε, των ε, ευρωπαϊκών περιφερειών. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Αντιπρόεδρο της Σουηδικής Κυβέρνησης για να μας μιλήσει εκ μέρους της Σουηδικής Προεδρίας. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι και μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών, κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που εκπροσωπώ εδώ μπροστά σας σήμερα τη Σουηδική Προεδρία κατά τα εγγένεια της φετινής ε, εβδομάδας Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Πόλεων. Η οργάνωση αυτή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να παραμείνω μαζί σας μέχρι ε, την ολοκλήρωση της εβδομάδας γιατί θα πρέπει να μεταβώ στη Σουηδία προκειμένου να παρουσιάσω ένα πρόγραμμα για τις ε, γυναίκες επιχειρηματίες. Γιατί ε, πιστεύω ότι και η δράση, η επιχειρηματική δράση των γυναικών θα αποτελέσει πηγή επιχειρηματικότητας ε, και ανάπτυξης περιφέρειες. Όταν ε, εκπρόσωποι όλων των ε, περιφερειών και των πόλων της Ένωσης συνέρχονται σε ένα κοινό χώρο για να συζητήσουν, θα υπάρξει αλλαγή, θα υπάρξει επικοδομητικός διάλογος και μια περιφερειακή απάντηση στις παγκόσμιες προκλήσεις. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία σας εδώ σε ό,τι αφορά την δυνατότητα να δώσουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση στις προκλήσεις αυτές, γιατί οι προκλήσεις έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα. Και η Ευρώπη, όπως και οι υπόλοιπε περιοχές του κόσμου, μαστίζονται από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δώσουμε μια παγκόσμια λύση στο πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών, γιατί είναι από τις πιο σημαντικές απειλές που αντιμετώπισε ποτέ η ανθρωπότητα. Οπότε είναι αυτονόητο ότι και η Ευρώπη και όλος ο κόσμος ε, έχουν συμφέρον ε, να ανταποκριθούν το συντομότερο δυνατό και με τον πιο επικοδομητικό τρόπο στις προκλήσεις αυτές. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις ε, σε διάφορα επίπεδα, σε ευρωπαϊκό αλλά και στο τοπικό και περιφερειακό ταυτόχρονα. Εγώ αισιοδοξώ ότι θα αντιμετωπίσουμε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα και το πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών και την επαναφορά στην οικονομική σταθερότητα έχουμε τώρα μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια οικονομία που θα εκμεταλλεύεται τις τεράστιες ευκαιρίες που υπάρχουν για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα και που θα προκύψουν από τις περιβαλλοντικές αλλαγές. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει την πρωτοκαθεδρία και να έχει ηγετικό ρόλο στη μεταμόρφωση της οικονομίας μας σε μια φιλοπεριβαλλοντική οικονομία. Και γι' αυτό θα πρέπει να υιοθετήσουμε καλοσχεδιασμένες πολιτικές, φιλόδοξους στόχους και να υποστηρίξουμε καινοτόμες τεχνολογίες που θα μπορέσουν να, αξιοποιήσουν το πλήρες δυναμικό της οικονομίας μας και να χρησιμοποιούν πιο ορθολογικά τους πόρους μας. Έτσι θα αυξήσουμε την ευημερία μας αλλά και την ανταγωνιστικότητά μας, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσουμε τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο και τον αντίκτυπο στις κλιματικές αλλαγές. Το ενεργειακό πακέτο για τις κλιματικές αλλαγές μας δίνει μια χρυσή ευκαιρία να αναλάβουμε έναν ηγετικό ρόλο στην ανέβρεση νέων λύσεων. Δεν μας ενδιαφέρει μια δεύτερη θέση. Θέλουμε την πρωτοκαθεδρία και γύρω στο 30% του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού Συνοχής αναμένεται να επενδυθεί στην πράσινη οικονομία. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί μάλιστα μέχρι το 2013. Χρειαζόμαστε φυσικά και τοπικές και περιφερειακές λύσει στις παγκόσμιες αλλαγέ. Γιατί οι Ευρωπαίοι πολίτες χρειάζονται περισσότερες θέσει απασχόλησης και καλύτερε, όχι μόνο στις πόλεις, αλλά και στην Ήπεθρο. Γι' αυτό και χώρε και οι περιοχέ θα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο από με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίω εφαρμόζοντα την πολιτική συνοχή. Το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να αναλάβει περισσότερε ευθύνε για την ανάπτυξη και στου συμμετοχή στους πόρους. Μια πιο ορθολογική χρήση των πόρων προϋποθέτει έναν εύρυθμο συντονισμό, μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων της τοπικής, περιφερειακής, εθνικής και ευρωπαϊκής. Ένας τρόπος για να το επιτύχουμε αυτό είναι να απλουστεύσουμε την εφαρμογή των ε, κοινοτικών ε, προγραμμάτων και της ε, εκταμίευσης των κοινοτικών κονδύλιων. Και αυτό προτείνουμε με την απλούστευση των διαρθρωτικών ταμείων. Και μάλιστα με βάση τη δική μου εμπειρία ως πολιτικού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά και ως διαχειρίστρια διαρθρωτικών προγραμμάτων, είμαι πεπισμένη θα πρέπει να απλουστευθεί η εφαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων όσο περισσότερο γίνεται. Και είμαι βεβαία ότι πολλοί θα συμφωνείτε μαζί μου και θα συμμερίζεστε την άποψή μου περί Βέβαια ταυτόχρονα συμφωνούμε ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να διαφυλάξουμε τις ε, θεμελιώδεις αρχές των διαρθρωτικών ταμείων και η χρήση τους θα πρέπει ε, να διέπεται από την αρχή της ορθολογικής και υπεύθυνης χρήσης των κοινοτικών κονδυλίων. Μία μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική συνοχή θα πρέπει να δώσει μια απάντηση στις παγκόσμιες αλλαγές. Και επίσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί σύνδεσμος μεταξύ της πολιτικής συνοχής και των στόχων της Λισαβόνας. Αυτή η στρατηγική προσέγγιση της πολιτικής συνοχής έχει συμβάλει αποτελεσματικά στη βελτίωση της απόδοσης των προγραμμάτων και στην εφαρμογή τους, ενώ ταυτόχρονα βελτίωσε τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων και την έκανε πιο αποτελεσματική. Γίνεται όλο και πιο σοφές ότι η ανταγωνιστικότητα και η ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτώνται από την πλήρη υλοποίηση και αξιοποίηση του δυναμικού των πολιτών της και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών. Οι καινοτόμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τμήμα της λύσης. Και ε, ο στόχος, ο Λισαβόνα, ότι θα πρέπει να έχουμε 60% ποσοστό απασχόληση για τις γυναίκες έχει σχεδόν πραγματοθεί. Και μάλιστα το ποσοστό αυτοαπασχόλησης των γυναικών δεν είναι τόσο ενθαρρυντικό. Δυστυχώς δεν αξιοποιείται πλήρως το δυναμικό των γυναικών και οι γνώσεις τους. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου το δυναμικό όλων των πολιτών όταν εξετάζουμε τις μελλοντικές ε, ευρωπαϊκές πολιτικές και όχι μόνο την, ε, την πολιτική συνοχής ή την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. Θα πρέπει βέβαια να αξιοποιήσουμε το ιδιαίτερο δυναμικό ανάπτυξης που έχει κάθε περιοχή χωριστά. Όλες αυτές οι ιδέες θα πρέπει να προσαρμοστούν με τρόπο που να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μέθοδοι που θα προσαρμόζονται στις ε, αδυναμίες και τα δυνατά σημεία της κάθε περιφέρειας. Και, και η πολιτική συνοχή θα πρέπει να προσανατολίζεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας. Είμαι πεπισμένη ότι θα πρέπει το πολιτικό αυτό μείγμα, το policy mix, να το προσαρμόσουμε στις ιδιάζουσες τοπικές και περιφερειακές συνθήκες. Γι' αυτό και η Σουηδική Προεδρία έχει θέσει ως ε, βασική της προτεραιότητα τη θέσπιση μακροπεριφερειακών στρατηγικών στο πρόγραμμα εργασιών της. Έχουμε φυσικά την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Βαλτική, που ευελπιστούμε ότι θα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τέλη του τρέχοντος ε, μήνα. Επίσης, ε, πιστεύουμε ότι μόνο και με μακροπεριφερειακή προσέγγιση μπορούμε να βρούμε απάντηση στις παγκόσμιες προκλήσεις. Και η προσέγγιση αυτή θα προσθεθεί στο πλωστάσιό μας για την αναζήτηση λύσεων. Και καλωσορίζω το έργο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία και μεταξύ των κρατών της περιοχής του Δούναβη. Η στρατηγική της Βαλτικής δεν θα πρέπει ε, να ειδωθεί ως αποδονωμένα. Θα μπορέσει να γίνει ε, πηγή έμπνευσης και για τις άλλες ε, περιοχές και να αξιοποιηθεί στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια θα έχουμε και πολλά σεμινάρια που θα εξετάζει αυτό το θέμα υπό διάφορες οπτικές πλευρές για τις επόμενες μέρες. Είναι σημαντική η ανταλλαγή απόψεων και παρουσίαση ιδεών σε τέτοιου είδους ε, διοργανώσεις και θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας από τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Γιατί αναγνωρίζουμε ότι η ποικιλία που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέσο για την αξιοποίηση του δυναμικού της Ένωσης. Η στρατηγική της Βαλτικής αναλύει κάποια προβλήματα που είναι ιδιαίτερα της ε, περιοχής αυτής, γιατί η Βαλτική είναι από τις πιο μολυσμένες θάλασσες του κόσμου και οι υποδομές στον ενεργειακό τομέα αντικατοπτρίζει τα πολιτικά χάσματα που υπάρχουν στην περιοχή αυτή. Και πιστεύουμε ότι χάρη στη συνεργασία τη διασυνοριακή και την διακλαδική θα βελτιωθεί η κατάσταση στη Βαλτική. Επίσης θέλουμε να βελτιώσουμε και το περιβάλλον στη Βαλτική θάλασσα και να ε, ενισχύσουμε την ολοκλήρωση και την ανταγωνιστικότητα στην περιοχή της Βαλτικής. Φυσικά θα πρέπει προηγουμένως να ενισχύσουμε και την εσωτερική αγορά και τις επενδύσεις στις υποδομές, προκειμένου να έρθει η περιοχή της Βαλτικής ε, πιο κοντά και κυριολεκτικά και όχι μόνο μεταφορικά στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να επενδύουμε σε καινοτομία και έρευνα όχι μόνο στο περιβάλλον και στην ενέργεια, αλλά σε όλους τους τομείς. Φυσικά κάτι τέτοιο προϋποθέτει νέους πόρους και νέα διοργάνωση, καλύτερη και πιο ορθολογική χρήση των υπαρχών των πόρων και πιο συντονισμένη δράση των προγραμμάτων. Θα θέλαμε οι πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις περιφέρειες ε, χωρίς επικάλυψη και χωρίς συμπληρωματικούς πόρους να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η περιοχή της Βαλτικής είναι μια μακροπεριοχή και έχει ε, πολύ ανταγωνιστική θέση σε πολλούς τομείς. Θα πρέπει να είναι μια γενική περιοχή αναγνωρισμένη για το περιβάλλον της, για το δυναμικό της στην έρευνα, για τις ε, ελκυστικές ε, συνθήκες εργασίας και πιστεύω ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις χρήζουν συνεργασίας και κοινή απάντησης. Θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί προς τις νέες ιδέες, χωρίς φυσικά να ξεχνούμε τα διδάγματα του παρελθόντος. Αυτή είναι η δική μου άποψη για τις απαντήσεις και τις λύσεις που θα χρειαστούμε, αλλά είμαι βεβαία ότι από την εβδομάδα των Open Days θα προκύψουν πολλές ιδέες και προτάσεις. Γιατί η ευρωπαϊκή λύση στα προβλήματα είναι το άθροισμα όλων των προτάσεων και λύσεων από το τοπικό και το περιφερειακό μέχρι το εθνικό. Μην ξεχνάτε ότι στους χαλεπούς καιρούς χρειαζόμαστε ισχυρή ηγεσία και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να βρίσκεται στην πρωτοκαθεδρία θα πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο για μια πράσινη οικονομία φιλοπεριβαλλοντική που θα λαμβάνει υπόψη και την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της κοινωνίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε Πρωθυπουργέ, ευχαριστούμε και τον ε, Πρόεδρο Μπαρόζο και την ε, εκπρόσωπο της Σουηδίας, την Πρωθυπουργό της Σουηδίας. Ξέρω ότι πρέπει να τρέξετε, να, προλάβετε μια πτήση, γιατί έχετε τόσα πολλά να κάνετε. Εμείς όμως θα μείνουμε σε αυτήν την αίθουσα, γιατί έχουμε τόσο σημαντικά πράγματα να συζητήσουμε. Τώρα εδώ με την βοήθεια του Τζάκι Ντέιβις από την, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής έχουμε τη διοργάνωση της υπόλοιπης ημέρας και ο Επίτροπος όμως Περιφερειακής Συνεργασίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Συνεργασίας του Ευρωκοινοβουλίου, όλοι είναι μαζί μας για τη συνέχεια της ημέρας μας, αλλά έχουμε και δύο προσκεκλημένους, τον Χέρμαν Χόρος, ο οποίος είναι εκπρόσωπος περιφέρειας της Ευρώπης και τον κύριο Άλβαρο, που είναι από την βασική κυβέρνηση της ε, Ισπανίας. Τους καλωσορίζουμε λοιπόν που βρισκόνται μεταξύ μας. Τζάκι, βρισκόμαστε στα χέρια σου για τα γεμάτα επαγγελματισμό. Thank Σας ευχαριστώ κυρία Χούμπνερ. Απλώς περιμένω τους προηγούμενους ομιλητές να αφήσουν την αίθουσα. Όπως είπε η κυρία Χούμπνερ, έχουμε ένα διτεκριμένο πάνελ σήμερα μαζί μας. Τους παρουσίασε ήδη, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω και εγώ λοιπόν. Έχουμε απλώς κάτι παραπάνω από μια ώρα για συζητήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να προλάβουμε όσο δυνατόν περισσότερες συνεισφορές να ακούσουμε και από εσά, αλλά να έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τις αποκρίσεις του Κοινοβουλίου. Εφόσον λοιπόν δεν έχουμε άλλους λόγους, ομιλίες, να περάσουμε απευθεία στις παρεμβάσεις σας, ερωτήσεις, και θα τα υποβάλλετε στο πάνελ, θα τους δώσουμε το λόγο και εάν ε, ε, μου επιτρέπετε να θυμίσω ότι όταν κάνετε τις ερωτήσεις σας να θυμάστε ότι πρέπει να υπάρχει χρόνος και για το πάνελ να απαντήσει. Λοιπόν, γιατί επειδή, ε, ε, ο, ο χρόνος πιέζει, και επειδή ανέφεραν οι προηγούμενοι ομιλητέ για την οικονομική κρίση, να στραφώ σε δύο από του συμμετέχοντε του πάνελ και να μα μιλήσουν για τι δικέ του εμπειρίε σχετικά με το θέμα αυτό. Κύριε Λόπε, η χώρα των Βάσκων είναι μια από τι πλουσιότερε περιοχέ στην Ισπανία και έχετε περάσει σοβαρέ προσπάθειε αναδιάρθρωση εσεί για να αντιμετωπίσετε τι προκλήσει τη παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Γνωρίζοντα ότι εργάζεστε σε αυτήν την παγκοσμιοποιημένη οικονομία, μπορεί η επιτυχία σα τελικά να σα κάνει και θύμα Πώς το αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό, πώς αντιμετωπίζετε αυτόν τον κίνδυνο. Καλησπέρα σας, καταρχήν. Και είμαι πεπισμένος πως όχι, γιατί στο παρελθόν δεν κάναμε προσπάθειες για να προσαρμοστούμε στις απαιτήσει μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Αυτό όμως σημαίνει ότι τώρα έχουμε μια καλύτερη θέση. Σήμερα βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση για να ανταποκριθούμε σε, σε απαιτήσει μια κρίση που και αυτή έχει παγκόσμιο χαρακτήρα. Και η έκθεση για τι περιφέρειες του 2020 τη Γενική Διεύθυνσης Περιφερειών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δείχνει ότι η χώρα των Βάσκων είναι η αυτόνομη περιοχή τη Ισπανίας που βρίσκεται σε καλύτερη θέση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων τη παγκοσμιοποίηση και των κλιματικών αλλαγών. Η χώρα των Βάσκων έχει λίγο παραπάνω από 2 εκατομμύρια κατοίκους πληθυσμό ε, που βρίσκονται σε 7.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα κατανεμημένοι. Και έχει ε, κατά κεφαλήνα 139 σχέση με το 100 που είναι ο κοινοτικό μέσος όρος. Έχουμε ποσοστό ενεργεία χαμηλότερο από το ισπανικό μέσο όρο και μεγάλο ποσοστό επιχειρηματικότητες, 26 και το ΑΕΠ ενώ το κοινοτικό είναι 18 και η παραγωγικότητα ε, έφτασε στο 132, δηλαδή 30 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το κοινοτικό μέσο όρο. Πώς εξηγούνται όλα αυτά, αυτές οι επιδόσεις της χώρας των Βάσκων. Η χώρα των Βάσκων είναι σίγουρα η περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανταγωνιστικότητας, γιατί έχουμε και σημαντικό ποσοστό αυτοδιοίκησης γιατί η χώρα των Βάσκων έχει μεγάλη εξουσία και μπορεί να εθετήσει τις πολιτικές πράξεις και τις νομοθετικές πράξεις που πειράζουν κατά το 90% τη ζωή των πολιτών. Αποφασίζουμε για την παιδεία, την υγεία, έχουμε δική μας αστυνομία, δικά μας μέσα μαζικής ενημέρωσης και έχουμε και μια άλλη ιδιαιτερότητα. Έχουμε οικονομικές εξουσίες ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις και για φορολογικά θέματα και οικονομικά. Οπότε έχουμε και πόρους που μας επιτρέπουν να υλοποιούμε τις αποφάσεις μας. Πριν από δύο εβδομάδες μόνο η κυβέρνηση των Βάσκων ενέκρινε ένα πακέτο, μια δέσμη μέτρων 400 ε, εκατομμύριων ευρώ που στόχο έχουν την καταπολέμηση των ε, άμεσων αποτελεσμάτων της κρίσης. Για παράδειγμα, θα ε, ενισχύσουμε κάποιες επενδύσεις σε δημόσια έργα και υποδομές που θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης αλλά και θα ε, δημιουργήσουν και προστιθέμενη αξία για το σύνολο της βασικής κοινωνίας και θα υποστηρίξουν το βιομηχανικό και επιχειρηματικό ιστό της χώρας των Βάσκων. Γιατί δεν θέλουμε ούτε μία βιώσιμη επιχείρηση της χώρας των Βάσκων να μην γονατίσει από την οικονομική κρίση. Γιατί άμα γονατίσει θα είναι δύσκολο να την ξανασηκώσουμε. Επίσης ε, η χώρα των Βάσκων ε, υποστηρίζει την καινοτομία, υποστηρίζει την διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. Επίσης ε, υπολογίζουμε στη μέθοδο που είναι καλύτερη για την καταπολέμηση της κρίσης και που είναι οι επενδύσεις στην παιδεία και την κατάρτιση, στην επιμόρφωση, στην κατάρτιση των νέων, στην, στον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων τους. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να διαμορφώσουμε και μια πιο αλληλέγγυα κοινωνία. Επίσης δίνουμε βάση στις πολιτικές κοινωνικών υπηρεσιών, γιατί δεν θέλουμε ούτε ένας πολίτης μας να υποστεί τις συνέπειες της κρίσης. Και σίγουρα θα πρέπει τα πιο αδύναμα στρώματα της κοινωνίας των Βάσκων να πληρώσουν τα σπασμένα για μια κρίση που δεν ήταν δική τους υπετιότητα. Ε, δεν θα πρέπει όμως να περιοριστούμε στο να δώσουμε κάποιες ε, απαντήσεις στα συμπτώματα της κρίσης. Θα πρέπει να θέσουμε ήδη τα θεμέλια για ένα νέο μοντέλο όχι μόνο οικονομικής ανάπτυξης αλλά διακυβέρνησης. Γιατί είπαμε ότι η κερδοσκοπία ήταν μία από τις αιτίες της κρίσης, η απορρίθμιση της αγοράς, το ελάχιστο βάρος του δημόσιου τομέα. Αυτή τη στιγμή όμως μπορούμε να τα θέσουμε όλα αυτά επιτάπητος και να βρούμε τα νέα θεμέλια και τις βάσεις για να καθορίσουμε χώρες και χώρους που θα είναι βιώσιμοι και αλληλέγγυοι μεταξύ τους. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε και νέα μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης που δεν θα στηρίζονται στην κερδοσκοπία, αλλά στην παραγωγικότητα και θα μπορούν να παράγουν, να πλούτο και να τον ανακατανέμουν με δικαιοσύνη. Μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο που θα είναι και βιώσιμο, αλλά και ποιοτικό και που θα συνδυάζει με ευφύ τρόπο τις παραδοσιακές με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα έχουμε και ένα νέο δημοσιονομικό και φορολογικό μοντέλο που θα είναι προοδευτικό, θα είναι δίκαιο, αλλά και αρκετό για να εφοδιάζει τις διοικήσεις με τα κονδύλια που χρειάζονται για να διεκπεραιώνουν το έργο τους. Και θέλουμε και ένα νέο μοντέλο ε, διαμόρφωσης και μετάδοσης της γνώσης και ένα νέο μοντέλο κοινωνικών, πολιτικών και υπηρεσιών γιατί η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι η πολιτική απασχόλησης και η αντιμετώπιση της ανεργίας. Βέβαια, πολλά από αυτά τα θέματα εκφεύγουν από τις δικές μας αρμοδιότητες, αλλά από τη δική μας τοπική και περιφερειακή εμπειρία καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αυτός ο συντονισμός είναι απαραίτητος για να διαμορφώσουμε ένα βιώσιμο και αλληλέγγυο μοντέλο. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε. Θίξατε μια πλειάδα θεμάτων. Πολλά ζητήματα τα οποία θα επανέλθουν στη συζήτηση. Να ρωτήσω τώρα και εσάς μια παρόμοια ερώτηση. Για αυτό που ονομάστηκε σαξονία της σιλικόνης με τόσες επενδύσεις στον τομέα των αυτοκινητοβιομηχανιών. Εσείς ε, πιστεύετε ότι η οικολογική προσέγγιση είναι μια διέξοδος από αυτή την οικονομική κρίση Πώς πιστεύετε ότι η επιτυχία σας μπορεί να εξακολουθήσει. Πιστεύετε ότι είστε βάλλοντες στις σημερινές συνθήκες. Ναι, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, βεβαίως ε, αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχουμε μία εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί όλες τις ε, περιφέρειες είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα σαφές μήνυμα για αυτές τις περιφέρειες. Να ξέρουν όλες τις περιφέρειες ότι αυτή τη στιγμή ασκείται μια περιφερειακή πολιτική και ότι η Λισαβόνα παίζει τον ρόλο που πρέπει να παίξει. Αυτό βέβαια ήταν ένα τμήμα της ερώτησης ε, και βεβαίως ξέρουμε ότι στην Δρέσδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά ε, προβλήματα σε σχέση με τις επιχειρήσεις, υπάρχουν μεμονωμένα προβλήματα ε, και υπάρχουν ε, προβλήματα σε σχέση με ορισμένες επιχειρήσεις, μικροηλεκτρονικής, αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά παρόλα αυτά έχουμε επιτύχει κάποια σταθερότητα. Καταφέραμε να επιτύχουμε μια ισορροπία, προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιες αντισταθμίσεις με μια συνεργασία που είχαμε με τις επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που είχαν διαφορετικούς προσανατολισμούς, προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε την οικονομία, να υπάρξει μια θεσμική συνεργασία και βεβαίως προσπαθήσαμε και για την φωτοβολταϊκή να δώσουμε μια νέα όθηση και βρισκόμαστε σε μια καλή κατάσταση, ικανοποιητική κατάσταση παρά την υπάρχουσα κρίση. Και βεβαίως και μπορούμε να πούμε ότι και ο τομέας των οικοδομών αυτή τη στιγμή είναι αρκετά ικανοποιητικός και όχι μόνο στη Δρέσδη αλλά και στην Ανατολική Γερμανία. Ξέρετε ότι πριν από 19 χρόνια ε, που έγινε η ειρηνική αυτή επανάσταση προσπαθήσαμε να βρούμε νέους τρόπους ανάπτυξης και ξέρουμε ότι οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο ευέλικτες στις αλλαγές που υπάρχουν, στις οικονομικές κρίσεις, υπάρχει μια αντίδραση και βεβαίως σήμερα μπορούμε να πούμε ότι τα καταφέραμε και έχουμε μια ικανοποιητική οικονομική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι αυτή η μεγάλη γερμανική πόλη κατάφερε να μην έχει χρέη και αυτό είναι ένα νόμιμο, και μια καινοτομία, κάτι το καινούριο. Πιστεύω ότι προσπαθήσαμε ε, να επιτύχουμε κάτι και δεν θέλουμε να είμαστε θύματα της ίδιας μας της επιτυχίας. Πιστεύουμε ότι η πόλη μας ε, τα κατάφερε, ιδιαίτερα στον τομέα της μικροελεκτρονικής. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν 40.000 ε, ε, απασχολούμενοι, υπάρχουν ε, πολλές επιχειρήσεις μικροηλεκτρονικής ε, και πραγματικά η μικροηλεκτρονική έχει πάρα πολύ αναπτυχθεί, έχουν δημιουργηθεί θέσεις απασχόλησης, υπάρχει καινοτομία, υπάρχει ένα πολύ ικανοποιητικό ποιοτικό επίπεδο, υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ της έρευνας, της οικονομίας και μεταξύ των αρχών. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της ε, περιφέρειάς μας και υπάρχει πραγματικά μια πάρα πολύ ικανοποιητική συνεργασία όλων των παραγόντων αυτής της περιφέρειας. Αυτή η ικανοποιητική συνεργασία ε, μπόρεσε να συνεισφέρει στο να επιτύχουμε μια τεχνολογική ανάπτυξη, μια ανάπτυξη των αγορών και μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι ε, και για τον τομέα της φωτοβολταϊκής και σε πολλούς άλλους τομείς στην, της προηγουμένης τεχνολογίας προσπαθήσαμε και καταφέραμε να έχουμε μια πολύ ικανοποιητική ανάπτυξη. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δέσμευση αυτής της περιφέρειας όλων των παραγόντων της και βεβαίως ε, είναι κάτι το οποίο μπορεί ε, να θεωρηθεί σαν μια πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί υπάρχει συνεργασία και με την Bundesregierung ε, και μπορούμε να πούμε ότι όλα μας ε, τα προγράμματα προωθήθηκαν και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε λοιπόν πολύ μεγάλες επιτυχίες στη Δρέστη ειδικότερα στον τομέα της ε, ανάπτυξης και της έρευνας. Η ανάπτυξή μας είναι πολύ ικανοποιητική. θα θέλαμε και πρέπει να πω ότι είμαστε ευγνώμονες γιατί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών υπήρξε μια καταφατική απάντηση από την πλευρά των Βρυξελών σε σχέση με την προηγμένη τεχνολογία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι υπάρχει στο μέλλον μια προοπτική, θα πρέπει να προωθήσουμε την καινοτόμο και προηγμένη τεχνολογία. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ ικανοποιητική κατάσταση και ξέρουμε ότι θα πρέπει ε, να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προηγμένη τεχνολογία από την οποία μπορούμε να περιμένουμε ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ακούσαμε λοιπόν τις εμπειρίες ανθρώπων που εργάζονται στο περιφερειακό επίπεδο. Και ένα από τα πράγματα που η σημερινή συνάντηση, τα Open Days, είναι ακριβώ αυτή η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, με αφορμή μάλιστα την κρίση. Σα ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερω. Ήθελα τώρα να στραφώ και πάλι στου ομιλητέ που είχαμε από το προηγούμενο μέρο τη συζήτηση για τι πολιτικέ συνέπειε ε, όλων των πολιτικών που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και από αυτά που ακούσαμε και από τους συμμετέχοντες του πάνελ και από τους προηγούμενους ομιλητές. Επίτροπε, να στραφώ σε εσά. Οι βραχυπρόθεσμες ανάγκες, η ταχύτερη υλοποίηση, πώς αντιμετωπίζονται αυτές τις ανάγκες τις πολύ άμεσες, πώς τις συνδυάζεται με τη διορατικότητα που χρειάζεται η ανάπτυξη πολιτικής ε, και προγραμματισμού των ε, ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά παντρεύονται με επιτυχία. Ε, Νομίζω η ανάγκη για ευελιξία δεν έχει να κάνει μόνο με τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες, αλλά ίσως ακόμη πιο πολύ και με τις μακροπρόθεσμες. Διότι σε έναν άμεσο ορίζοντα είναι πολύ εύκολο κανείς να επιλύσει ένα πρόβλημα ε, με έναν τρόπο πρόχειρο. Όμως ε, για να δει κανείς έναν μακροπρόθεσμο ορίζοντα πρέπει να δει κάποιες ε, τάσεις διαρκείας. Αυτό το ανέφερε και ο Πρόεδρος όταν ε, μίλησε για την ανάγκη οι περιφέρειες να συμμετέχουν ενεργότερα στη διαδικασία τη Λισαβόνας. Να ακούμε τις ιδέες των περιφερειών και τις καινοτόμε προσεγγίσεις τους. Ανέφερε την έλλειψη ευθύνη και ιδιοκτησία για τη στρατηγική τη Λισαβόνα, κανεί δεν φαίνεται να είναι ακριβώ υπεύθυνο για αυτήν και αυτό λείπει. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικέ προσεγγίσει ανάλογα με τα κράτη-μέλη, τι περιφέρειε και τι μεγαλύτερε περιφέρειε, όπω η στρατηγική τη Βαλτική θάλασσα. Άρα η ανάγκη για περισσότερη ευελιξία δεν αναφέρεται μόνο στι βραχυπρόθεσμε ανάγκε, αλλά και στι μακροπρόθεσμε. Και τι να πω εδώ. Να πω ότι προφανώς θα ήταν ε, κάπως ε, Ριψοκίνδυνο να μην ε, συμφωνήσω μαζί σας, αλλά συμφωνώ γιατί είναι και αλήθεια αυτό που λέτε. Ωστόσο, θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα και θα έλεγα ότι χρειάζεται περισσότερη συμμετοχή των περιφερειών στον σχεδιασμό της δαπάνης, των δαπανών και της χρήσης των πόρων, αλλά και μεγαλύτερη προσπάθεια για την εκδίπλωση των ικανοτήτων τους. Δηλαδή θα πρέπει, ε, αν θέλετε περισσότερη εξουσία ως περιφέρειες, να είστε και περισσότερο υπόλογοι βεβαίως και να μπορείτε να εξηγήσετε τις, επιδο... τις επιδόσεις σας, την ε, δημοσιονομική σας, την οικονομική σας πειθαρχία να μπορείτε να αποδείξετε. Οι πόροι και η διαχείριση των πόρων δεν είναι απαλλαγμένοι από ατασταλίες. Περισσότερη λοιπόν εξουσία στις περιφέρειες, αλλά και περισσότερη ευθύνη ταυτόχρονα. Και ανάληψη ευθυνών για την επίτευξη καλών επιδόσεων. Ευχαριστούμε πραγματικά. Κυρία Χούμπνερ, όταν είσαστε επίτροπο για την περιφερειακή ανάπτυξη και εσεί αναλάβατε πρωτοβουλία, όπω είπαν και άλλοι ομιλητέ, αναλάβατε μέτρα για να απλουστεύσετε τι διαδικασίε στήριξη των περιφερειών, ιδίω από την έναρξη τη οικονομική κρίση. Έχοντα κατά νου λοιπόν αυτό που μόλι μα είπε ο επίτροπο, για την ανάγκη να υπάρχει ισορροπία μεταξύ υπολόγου ευθύνη και ανάπτυξη, πιστεύετε ότι έχουν γίνει αρκετά για να γίνει πιο ευέλικτο το σύστημα, για να υπάρξει απλούστευση, ή υπάρχουν περαιτέρω βήματα τα οποία υπό τη νέα σα ιδιότητα θα μπορούσατε να προωθήσετε στο Ευρωκοινοβούλιο. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε μια μακροπρόθεσμη και μακροχρόνια διαδικασία με την απλοποίηση αλλά και με τις συστάσεις ε, για πολλές νομοθετικές αλλαγές. Και οι παλιότεροι από σας ε, θα θυμάστε πιο πολέμαχοι ότι εντοπίσαμε την ανάγκη απλοποίησης ε, τη ε, περιφερειακή πολιτική. Αυτό το είπαμε πριν από πολλά χρόνια. Μόνο όμω όταν μα χτύπησε η κρίση, όταν χτύπησε η κρίση την πραγματική οικονομία, ξαφνικά συμφώνησαν όλα τα κοινοτικά θεσμικά όργανα ότι όντω χρειάζεται απλοποίηση και ε, ξεκίνησε επιτέλου αυτή η διαδικασία. Από την άποψη αυτή δηλαδή η κρίση δημιούργησε την ευκαιρία αυτή για την απλοποίηση. Η περιφερειακή πολιτική δεν απλουστεύτηκε μόνο, δεν είναι ότι έγινε μόνο κάποια ελαστικοποίησή της αλλά έγινε καλύτερος προσανατολισμός των επενδύσεων στις πιο ευφυείς ε, ε, προτάσεις και η περιφερειακή αυτή είναι εκφύσεως πολιτική μακροπρόθεσμων επενδύσεων, διαρθρωτικών επενδύσεων. Γι' αυτό και υπάρχουν προγράμματα που στηρίζονται στην αναπτυξιακή στρατηγική, την τοπική, περιφερειακή και εθνική αναπτυξιακή στρατηγική. Ο ίδιος ο σχεδιασμός λοιπόν της πολιτικής ε, την έκανε κατάλληλη για να ανταποκριθεί στη κρίση. Γιατί δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την κρίση ξεχωριστά από την βιώσιμη ανάπτυξη. Γιατί η κρίση αυτή είναι κέρδη αρθρωτική και θα εξέλθουμε από αυτή μόνο αν εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες της και προβούμε στις κατάλληλες επενδύσεις ε, για τις οποίες μας μίλησε ο κύριο πρόεδρος Πάτσι Λόπες για τις προσπάθειες που έκανε η βασική κυβέρνηση. Τα τελευταία χρόνια καταλήξαμε σε προτεραιότητες που θα μας επιτρέψουν ε, να δώσουμε απαντήσεις στην κρίση και που χρησιμοποιούν μια διαρθρωτική και στρατηγική προσέγγιση και προσπαθούν ε, να προσελκύσουν και ιδιωτικέ επενδύσει και όχι να τι απομακρύνουν. Επίση, υπάρχει ένα χρηματοπιστωτικό μέσο που είναι μακροπρόθεσμο και θα μα βοηθήσει να εξέλθουμε από την κρίση. Γιατί η κρίση είναι και κρίση των επενδυτικών ε, ταμείων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι τράπεζε ακόμη προσπαθούν ε, να διορθώσουν του ισολογισμού του και να εξηγιάνουν τα οικονομικά τους σε σχέση με τις εγγύησεις που έδωσαν. Νομίζω ότι η περιφερειακή πολιτική θα είναι μία από τις πολιτικές εξόδου από την οικονομική κρίση. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος. Είπατε πριν από λίγο, κύριε Πρόεδρε, ότι κανείς δεν ξεκινάει να χτίσει σπίτι από την οροφή. Η προσοχή όμω του κοινού και το μέσο μαζική ενημέρωση επικεντρώθηκε σε επίπεδο οροφής, σε επίπεδο κορυφής και ιδιαίτερα διάσκεψη κορυφής σε G20 στο Pittsburgh. αναμένεται και η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για το περιβάλλον. Υπάρχει όμως συντονισμός και στις πιο χαμηλές βαθμίδες γιατί οι περιφέρειες είναι αυτές που υλοποιούν και δίνουν σάρκα και οστά στα προγράμματα. Έχουν ανάμειξη στην ε, συνολική διαδικασία και οι περιφέρειες. Ναι, υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης ό,τι αφορά την ανάπτυξη των δήμων και κοινοτήτων, των περιφερειών στην παγκόσμια λύση. Δυστυχώς η προσέγγιση όμως από κυριαρχεί είναι από την κορυφή προς τη βάση αντί να είναι η αντίστροφη. Και εξετάζοντας τα πράγματα βραχυπρόθεσμα, διαπιστώνουμε ότι η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση έχει πληγεί τα μάλα από την χρηματοπιστωτική κρίση. Ένα τρίτο όλων των κρατικών δαπανών ε, δίνονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και δύο τρίτα των συνολικών επενδύσεων της Ένωσης ε, γίνονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Θέλετε και άλλα παραδείγματα για να αντιληφθείτε ότι μόνο και μόνο για να υλοποιήσουμε τους συνολικούς μας στόχους, τους παγκόσμιους στόχους, χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό και συνεργασία των θεσμικών οργάνων με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Πιστεύω ότι για να πραγματώσουμε όλους αυτούς τους στόχους θα πρέπει, όπως είπα και προηγουμένως, να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όπου η πολιτική συνοχή θα προσανατολίζεται προς τους στόχους της. Η πολιτική αυτή όμως θα πρέπει να καλύπτει όλες τις περιοχές. Δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα κατακαιρματισμού των προγραμμάτων της Ένωσης. Θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι νέες, οι νέες γραμμές της στρατηγικής Λισαβόνας και μετά το 2010, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε διασύνδεση και με τα προηγούμενα προγράμματα. Μην ξεχνάτε ότι ένα από τα κεντρικά θέματα το, της εβδομάδας αυτής θα είναι η καινοτομία. Πού βρίσκεται η καινοτομία? Στους πόλους αριστείας μας, στα κέντρα αριστείας και στα πανεπιστήμια. Και εκεί πραγματικά υπάρχει πρόοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και από θέματα προϋπολογισμού και αναθεώρησης των δημοσιονομικών προοπτικών οι επιτροπές περιφερειών ε, πιστεύουν ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα για να φτάσει η πρόοδος προς τους πολίτες. Δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε σε θεσμικό μόνο πλαίσιο. Βλέπω τον καλό μου φίλο κύριο Βανίστερ Ρόι και τους άλλους ευρωβουλευτές και χαιρόμαστε που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποκτήσει περισσότερες εξουσίες μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας φαίνεται ότι αρχίζει και γίνεται πιο συγκροτημένο το θεσμικό οικοδόμημα. Και όταν λέμε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι χρειάζονται εταιρική σχέση, δεν αντιβαίνουμε στη συνθήκη και όταν ζητούμε πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, το αντίθετο. Μην ξεχνάτε τι έκανε η Επιτροπή Περιφερειών τα προηγούμενα χρόνια και η Επιτροπή η Κοινωνική και η Οικονομική Επιτροπή επιζητούσαν έμπρακτες λύσεις, ρεαλιστικές λύσεις. Και το λέω συνεχώς στον πρόεδρο Μπαρόζο. Αν λάβετε υπόψη τις τοπικές και περιφερειακές προτάσεις θα είστε πιο αποτελεσματικοί και πιο αποδοτικοί. Είδαμε σε ευρωεκλογές ότι μόνο το 43% των ψηφοφόρων πήγαν στις κάλπες για να ψηφίσουν. Αυτό είναι το μήνυμα ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν να συμμετέχουν αλλά επίση ίσης με τα θεσμικά όργανα και είναι κατά των διαπληκτισμών και του θεσμικού πολέμου. Καλώ. Θα ακούσουμε ορισμένε ερωτήσει από το κρατήριο. Θα είμαι όμω πολύ αυστηρή στην κατανομή του χρόνου, γιατί ήδη πολλοί ε, ζήτησαν το λόγο και φαντάζομαι και άλλοι θα τον θέλουν. Παρακαλώ οι ερωτήσεις να είναι μονόλεπτες γιατί αν παραβεί κάποιο το χρόνο του θα πάρω το σφυρί από την πρόεδρο Χίμπνερ. Ελπίζω να μην χρειαστεί. Θα ήθελα παρακαλώ όλοι, όλοι όσοι θέλουν να, να θέσουν ερωτήσεις να σηκώσουν το χέρι τους για να ξέρω πόσοι ομιλητές θα είναι στο κατάλογο. Θα παίρνω έναν από το κατάλογο που έχω μπροστά μου και ένα από το ακροατήριο. Κυρία Μερσέδες Πρέστο από την, την περιοχή του Πιεμόντε. Ευχαριστώ. Όπως αναφέρθηκε πριν, υπάρχει αυτή η οικονομική κρίση και ε, βεβαίως απευθύνονται οι πολίτες πρώτα στους ε, ηθήνοντες της ε, περιφερειάς τους και στην δική μου περιφέρεια έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα για να μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, και βεβαίως για να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες αυτή τη στιγμή της κρίσης. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να εμβαθύνει ο Επίτροπος σχετικά με το θέμα της ευελιξίας των μέτρων συγχρηματοδότησης σε σχέση με το Κοινωνικό Ευρωπαϊκό Ταμείο. Και αυτή τη στιγμή προφανώς είναι πολύ σημαντική αυτή η προσφυγή δυνατότητα ε, για τους άνεργους και για τη δημιουργία βεβαίως νέων θέσεων εργασίας ιδιαίτερα στο θέμα της πράσινης οικονομίας στον τομέα της πράσινης οικονομίας. Θα ήθελα λοιπόν ε, να θέσω αυτή την ερώτηση και να δούμε πόσο μπορούμε να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα ε, στην διασυνορική συνεργασία, στη συνεργασία μεταξύ των περιφερειών. Υπάρχουν πολλές ε, ε, καθυστερήσεις, θα πρέπει να υπάρξει μία συνεργασία και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να υπάρξει μία συγκεκριμένη βελτίωση στην λειτουργικότητα. Θα πρέπει να υπάρξει μία επιτάχυνση γιατί αυτός ο τομέας είναι εξαιρετικά σημαντικός για μας. Καλώς κάποιος από το ακροτήριο που δεν, ε, ε, δεν έχει εγγραφεί στον κατάλογο των αγορητών. Ε, Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Φρανσίσκο Δελατόρε και είμαι ο δήμαρχος της Μάλαγα, της περιοχής της Ανταλουσίας με περίπου 600.000 πληθυσμό. Είμαστε τέσσερις Ισπανοί ε, δήμαρχοι που εκπροσωπούμε τους 8.000 δήμους και κοινότητες της Ισπανίας στην Επιτροπή των Περιφερειών. Για να αντιμετωπίσουμε την κρίση πιστεύω ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε πλήρως την αρχή της επικουρικότητας. Ορισμένες χώρες όπως η Ισπανία δεν έχουν αξιοποιήσει πλήρω την αρχή τη επικουρικότητα. Στην Ισπανία από το 1978 μέχρι σήμερα, δηλαδή θα ολοκληρώσουμε 30 χρόνια το Δεκέμβριο, έχουμε εγκρίνει το ψήφισμά μα και έχουμε εφαρμόσει ένα σύστημα αυτόνομης αποκέντρωσης πολύ αποτελεσματικό και ο πρόεδρος Πατσιλόπες ε, αποτελεί ένα υπόδειγμα αυτής της περιφερειακής αυτονομίας. Εδώ και 30 χρόνια όμως ε, δεν έχουμε καμία προσπάθεια για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων από το κεντρικό στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Γιατί οι αυτονομίες έχουν λάβει κάποιες εξουσίες αλλά δεν τις έχουν μεταφέρει καλά στις περιφέρειες και τους δήμους οι ψηφοφόροι μας ζητούν από τους δημάρχους ε, απτές κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης. Στην Ανταλουσία έχουμε 25 27% ανεργία, όχι όπως στη χώρα των Βάσκων. Υψηλό ποσοστό ανεργίας. Δεν λέω ότι η μόνη λύση θα προκύψει από την εφαρμογή της αρχής επικουρικότητας. Θέλουμε ανταγωνιστικότητα σε θέματα καινοτομίας, ε, γνώσης, έρευνας. Αλλά θα πρέπει η κοινωνική πολιτική, η πολιτική απασχόληση εφαρμόζονται από τους Δήμους και τις κοινότητες. Έχουμε την ε, ε οργανισμό, τον τοπικό οργανισμό περιβάλλοντος. Έχουμε, είχαμε πρωτοστατήσει σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Πιστεύουμε ότι για όλα αυτά έχουμε υποχρέωση να αναλάβουμε δράση, γιατί μα το ζητά ο ίδιο ο κόσμο. Θα πρέπει οι Δήμοι και οι κοινότητε να δώσουν μάχη για να εφαρμοστεί πλήρω η αρχή τη επικουρικότητα παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε έπειτα τι απόψει των μελών του πάνελ. Και τώρα, η Κωνσταντ Κλέρ. Ευχαριστώ. Εδώ είμαι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή την Περιφερειακή Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στην Επιτροπή. Πόσα εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Τι έγινε, τι συγκεκριμένες αλλαγές υπάρχουν, κατά πόσο είναι λειτουργικά αυτά τα προγράμματα, πόσο κατά πόσο εφαρμόστηκαν αυτά τα προγράμματα. Παραδείγματος χάρη στο θέμα της κοινωνικής κατοικίας. Πόσες, ε, πόσες κατοικίες δόθηκαν αυτή τη στιγμή διατέθηκαν στους πολίτες. Ε, ακούσαμε τι έγινε στη Δρέσδη, ακούσαμε τι έγινε στη χώρα των Βάσκων. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω ότι και οι Βάσκοι και οι Δρέσδη είναι ικανοποιημένες ε, Πρόκειται για δύο περιφέρειες οι οποίες ε, μπορέσαν μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής ε, να προκόψουν, ε, να περάσουν σε ένα στάδιο ανάπτυξης, ανάκαμψης και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα πρέπει βεβαίως να υπάρχει μια μεγαλύτερη συμμετοχή στις επόμενες ευρωεκλογές από αυτή που είχαμε την τελευταία φορά θα έπρεπε ίσως να υπάρχει μια καλύτερη διαφήμιση, μια καλύτερη ενημέρωση θα πρέπει να ξέρουν οι πολίτες τι κάνουμε για αυτούς και αυτό δεν νομίζω ότι είναι αρκετά γνωστό. Ευχαριστώ. Θα δώσω την ευκαιρία στους δύο πάνελιστ να σας ανταποδώσουν τις τα ευγενικά σα λόγια, αλλά προηγουμένω σα ακούσουμε ακόμα κάποιε ερωτήσει. Κάποιο από το ακρατήριο που να μην είχε πει εκ των προτέρων ότι θέλει να παρέμβει, εκεί πίσω-πίσω, στο βάθο. Ε, βάζω ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό για εμάς που επενδύσαμε σε, ε, να παράγουμε αγροτικά προϊόντα και υπάρχει κίνδυνος πραγματικά όχι μόνο σε εμάς στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης επενδύσεις οι οποίες έγιναν με επιδοτούμενα προγράμματα από Λίντερ για το μέτρο 2.1 και άλλα προγράμματα ε, έχω ανταλλάξει απόψεις και με Ιταλούς και με Ισπανούς και με άλλους συναδέρφους κινδυνεύουμε να κλείσουν αυτές οι επενδύσεις και λέω ε, κάτι και ζητάω κάτι σοβαρό πώς δίνονται κίνητρα για να αγοράζονται ηλεκτρονικά μέσα ή οτιδήποτε σε καταναλωτές γιατί να μην δίνεται ένα κίνητρο στον καταναλωτή να αγοράζει προϊόντα βιολογικά και προϊόντα που παράγονται στη Μεσόγειο, στα κράτη τα δικά μας. Και καταναλώνουν προϊόντα οι Ευρωπαίοι, τα οποία εγώ τα ονομάζω πλαστικές τροφές, τα οποία έρχονται από χώρε που δεν είναι μέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Αυτό θέλω μια απάντηση σε αυτό. Okay. Thank you very much indeed. Um, Σας ευχαριστούμε. Κλάου Κλάκλας από το Δημοτικό Συμβούλιο της Λίβερ Έχει φύγει κυρία. Από το Συμβούλιο του Κέρι Κάουντι. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της ομάδας μας θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους και να σας ευχαριστήσω για τη διοργάνωση και ως Ιρλανδός θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια μετά την βροντερή φωνή της Ιρλανδικής ετοιμιγωρίας το περασμένο Σαββατοκύριακο. Αυτό δείχνει ότι οι Ιρλανδοί θέλουν να βρίσκονται στην καρδιά της Ευρώπης και θεωρούν ότι το μέλλον τους ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε δύσκολη εκλογική εκστρατεία δημοψηφίσματος στην ε, ε, Ιρλανδία και υπήρξε ένα τεράστιο έλλειμμα πληροφόρησης και ενημέρωσης. Ε, και ο μέσος Ιρλανδός πολιτής δεν είχε γνώση της κατάστασης. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταγράψει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολιτών σε όλες τις πόλεις και την περιφέρεια. Αν κάτι διδαχθήκαμε από την Ιρλανδική εμπειρία, αυτό θα πρέπει να είναι ότι όταν οι Ιρλανδοί δεν γνώριζαν τα πράγματα, ψήφισαν όχι. Όταν ενημερώθηκαν, έδωσαν μαζικά την έγκρισή τους και ψήφισαν ναι στη Λισαβόνα. Υπήρχε ένα τεράστιο ε, έλλειμμα πληροφόρησης προηγουμένως στην Ιρλανδία για το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς επηρεάζονται οι πολίτες. Οι πολίτες δεν ήταν αρκετά πληροφορημένοι για τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή η άγνοια οδήγησε σε μια αρνητική εντύπωση των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν, αν συμφωνούμε ότι υπάρχει ε, έλλειμμα ενημέρωσης ε, και συμφωνούμε προ τη διάγνωση τι σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πράξει προκειμένου να γεφυρώσει αυτό το χάσμα της ενημέρωσης για τους πολίτες. Φαντάζομαι παρόμοιε πορείες έχουν και άλλοι συνάδελφοι. Ο κύριο Κέλλη, Ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ. Έρχομαι από την ίδια περιοχή με τον προηγούμενο ομιλητή τον κύριο Ντονάχιο και είμαι βουλευτή. Ευχαριστώ τον κύριο Βάντεμπραντ και τον κύριο Μπαρόζο για τα θαυμάσια σχόλιά του. Και οι δύο είπαν ευχαριστούμε Ιρλανδία. Εμεί από τη μεριά μα θέλουμε να πούμε ευχαριστούμε Ευρώπη. διότι θα ήταν πραγματικά παράδεκτο να απορριφθεί και πάλι η συνθήκη τη Λισαβόνα και κατά την εκστρατεία για το δημοψήφισμα, ο κύριος Μπαρόζ επισκέφθηκε το Λιμερίκ και είπε ότι το Ταμείο για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση θα αποδεσμεύσει κονδύλια για τους εργαζόμενους εκεί που έχουν χάσει τις δουλειέ τους. Να λοιπόν τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ιρλανδία. Πάντως, για τον νότο της Ιρλανδία να πω ότι δυστυχώς έχουμε προβλήματα φτώχεια αλλά έχουμε μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε μια αρκετά πιο ευημερούσα περιοχή, ακριβώ χάρη στη στήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κρίση βέβαια μα έχει χτυπήσει, μα μαστίζει χωρί ήκτο και έχουμε και πάλι καθυστέρηση στην οικονομική ανάπτυξη. Η Επιτροπή λοιπόν πρόκειται να αναθεωρήσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας για στήριξη από τα Ταμεία Συνοχής όπως για την Ιρλανδία λόγου χάρη. Σας ευχαριστώ. Θα επανέλθω τώρα στο πάνελ και μετά θα έχουμε και πάλι γύρω ερωτήσεων. Δεν ξέρω ποιοι ακριβώς θέλουν να πάρουν το λόγο πριν απαντήσουν οι πάνελιστ. Ας ακούσουμε όμως και πραγματικά καλό, κάντε και μια μικρή επιλογή μεταξύ των ερωτήσεων που ακούσατε. Απαντήστε σε αυτά που θέλετε για να μπορέσουμε να ξανακούσουμε ερωτήσεις. Τώρα, ο πρόεδρος της χώρας των Βάσκων, η δήμαρχος, Θέλετε να απαντήσετε σε κάτι από όλα αυτά που ακούσατε, να κάνετε σχόλια. Θα απαντήσω σε δύο ερωτήσεις. Είναι προφανές ότι η ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιφέρειές μας είχε κεφαλαιόδη σημασία για την οικονομική μας πρόοδο στη δεκαετία του 80, γιατί τότε η χώρα των Βάσκων υπέστη δινή κρίση και κατάφερε να εξέλθει από αυτή με την αλλαγή του παραγωγικού ιστού, με την ε, διαφοροποίηση της ε, βιομηχανίας και με την ενίσχυση των περιοχών χάρη σε κοινοτικά κονδύλια. Και η βασική κοινωνία είναι φιλοευρωπαϊκή, γιατί μεταξύ άλλων ε, η διεισόμαση διαπίστωσε ότι μια Ευρωπαϊκή Ένωση εφοδιασμένη με πόρους που θα τους διοχετεύσει εκεί που χρειάζονται είναι απολύτως απαραίτητη για όλους. Θα πρέπει βέβαια να έχουμε επίγνωση των σχετικά μικρών διαστάσεων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Γι' αυτό και τα ισχνά κονδύλια που υπάρχουν θα πρέπει να διατίθενται στις περιοχές που πραγματικά θα επιφέρουν θέμενη αξία και θα ενισχύσουν μειονεκτικούς τομείς και περιοχές. Γιατί εκεί θα φανεί η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των αναγκών και των προβλημάτων των πολιτών. Και εκεί θα πρέπει να ε, εστιαστούν οι δράσεις και τα κονδύλια της Ένωσης, ιδιαίτερα τα διαφορετικά, δηλαδή στις πιο μειονεκτικές περιοχές, τα πιο μειονεκτικά στρώματα του πληθυσμού και στις διασυνοριακές ε, προσπάθειες και προγράμματα προκειμένου να διαμορφωθεί μια πεδία συνεργασίας και αλληλεγγύης. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια του Δημάρχου της Μάλαγας, εγώ είμαι υπέρμαχος της επικουρικότητας στην πολιτική και πιστεύω ότι θα πρέπει με ορθολογικότητα και κοινή λογική να εφαρμόσουμε την επικουρικότητα. Μάλιστα, μια κατανομή των πολιτικών αρμοδιοτήτων θα πρέπει να υπακούει στην κοινή λογική και στην ανάγκη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Δυστυχώ η κατάσταση που περιγράψατε δεν είναι ομοιόμορφη σε όλη την Ένωση. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ε, δήμοι που δεν έχουν καμία αρμοδιότητα, ε, που δεν έχουν ε, λάβει εξουσίες από τις αυτονομίες. Παρ' αυτά, είναι αλήθεια ότι η Δήμη είναι το πρώτο παράθυρο, η πρώτη θηρίδα στην οποία αποτείνεται ο πολίτης όταν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Και θα πρέπει οι κυβερνήσεις ε, και σε κρατικό επίπεδο και σε επίπεδο αυτονομίας να εξασφαλίζουν πόρους στους Δήμους για να μπορέσουν να διεκπαιρεώσουν το έργο τους. Και μάλιστα αυτό να γίνει ε, πηγόντως γιατί η κατάσταση πραγματικά είναι επίγουσα. Κυρία Δήμαρχος της Δρέσδης. Ναι. Καταρχήν, θα ήθελα να δώσω μια απάντηση στο θέμα των περιφερειών στην Ευρώπη. Βεβαίως ε, υπάρχουν τομείς στους οποίους δεν έχω ε, αρμοδιότητα. Ε, πρόκειται για την περιοχή που είναι κοντά στην Τσεχία και στην Πολωνία και για, πρόκειται βέβαια για την διασυνοριακή ε, συνεργασία. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας παρέχονται από αυτή τη διασυνοριακή συνεργασία και βεβαίως υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες ε, συνεργάζονται και οι οποίες προέρχονται από και από τις τρεις αυτές χώρες. Πρόκειται λοιπόν για μια ε, πολύ ενδιαφέρουσα συναστρία. Υπάρχουν τέτοιες ε, ε, περιφέρειες οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ότι αποτελούν ένα μοντέλο, ένα υπόδειγμα. Ο συνάδελφος από την Μάλαγα αναφέρθηκε σε αυτά που και εγώ ήδη έχω πει ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να μπορέσουμε πραγματικά να εφαρμόσουμε τις πολιτικές μας και αυτό εξαρτάται από όλους μας, από τον καθένα μας, από τους πολίτες. Βεβαίως υπάρχει το θέμα των αρμοδιοτήτων. Εμείς στη Γερμανία, στην περιοχή του Ζάξεν, πρέπει να πω ότι έχουμε επιτύχει πάρα πολλά πράγματα και στον τομέα των αρμοδιοτήτων ε, Υπάρχει δηλαδή μεγάλη ανεξαρτησία και των Λέντερ και συνεργασία με την Bundesregierung. Ε, θα ήθελα να πω κύριε που, ότι φυσικά συμφωνώ με την άποψή σας αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα με μονομένα άτομα να προωθήσουν αυτές τις απόψεις με τον τρόπο που το ζητήσατε. Υπάρχουν άλλες δυνατότητες οι οποίες μας παρέχονται και εδώ δεν υπάρχει καμία αντίφαση με τις απόψεις που ήδη εσείς διατυπώσατε ε, νομίζω ότι και στην Γερμανία και στο Ζάξεν μπορούμε να πούμε ότι πετύχαμε πάρα πολλά πράγματα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής συνεργασίας και σε θέματα διαρθρωτικών πολιτικών αλλά και σε άλλους τομείς. Βεβαίω βεβαίως ε, θα ήθελα να δώσω και εγώ νερό στο μήλο σας ε, και να πω ότι θα πρέπει να κινηθούμε με μεγαλύτερη ταχύτητα να ε, μπορέσουμε πραγματικά να απλοποιήσουμε και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Είναι ένα πρόβλημα. Υπάρχει το πρόβλημα της ε, συνεργασίας, του συντονισμού, του δημόσιου τομέα. Νομίζω λοιπόν ότι σε γενικές γραμμές υπάρχει βελτίωση. Πάμε καλά. Ευχαριστούμε. Επίτροπε, υπήρχαν ε, τουλάχιστον δύο-τρία ερωτήματα που αναφέρονταν σε εσά για το έλλειμμα πληροφοριών αλλά και για την συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και πώς ε, μπορούν να είναι επιλέξιμε περιφέρειε για τη συγχρηματοδότηση και πόσο δυσκολεύονται με αυτό το σύστημα το σημερινό. Συγκεκριμένα ερωτήματα. Ναι, όντω είναι πολύ συγκεκριμένα και η Επιτροπή έχει προτείνει δύο πακέτα με σκοπό την απλούστευση και την διευκόλυνση της χρηματοδότησης ε, των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το πρώτο επειδή είχε εγκριθεί, έδωσε τη δυνατότητα για προκαταβολές, πληρωμές δηλαδή εκ των προτέρων, ταχύτερα ήδη τον Απρίλιο φέτος, 6,25 εκατομμύρια ευρώ αποδεσμεύτηκαν και μεταφέρθηκαν στα κράτη. Άλλες διατάξεις αυτού του πακέτου ήταν ε, η τροποποίηση των επιχειρησιακών, ε, των λειτουργικών προγραμμάτων, ταχύτερη έγκριση των ε, προγραμμάτων και η ταχύτερη αποδέσμευση πόρων, η αύξηση του κατοφλίου για την επιλογή προγραμμάτων, τα οποία πρόκειται να ελέγχονται στη συνέχεια με τρόπο διαφορετικό ως 50 δις, λέει ο ευρώ, όλα αυτά πλουστεύουν την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής. Η Επιτροπή έχει κάνει και άλλη μια πρόταση για 100% συγχρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Όμως η πρόταση αυτή επικρίθηκε ιδιαίτερως από το κρατημέλη. Σήμερα λοιπόν αναζητούμε εναλλακτικέ λύσεις. Αυτό αφορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα διαφορετικά. Και πολύ σύντομα για το έλλειμμα πληροφόρησης που αναφέρθηκε. Η Επιτροπή βεβαίως κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν μπορεί να πάρει τις ευθύνες των κρατών μελών, των κυβερνήσεων, των τοπικών αρχών, των μέσων μαζικής επικοινωνίας, των δημοσιογράφων, των προσωπικότητων και των δημόσιων προσώπων. Η οικοδόμηση της Ευρώπης δεν είναι ένα καθήκον της Επιτροπής μόνης, είναι ένα καθήκον συλλογικό όλων μας. Συμφωνούμε ότι υπάρχει έλλειμμα λοιπόν ενημέρωση, όμω αυτό πρέπει να καλυφθεί από πολλού παράγοντε, όχι μόνο από την Επιτροπή. Και είναι ένα ζήτημα αυτό που έχει να κάνει και με τα κριτήρια επιλεξιμότητα. Θα αλλάξουν, μα ρωτάτε. Όχι, δεν υπάρχει μυστική συμφωνία μεταξύ Επιτροπή και Ιρλανδία. Θα διατηρηθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητα, τουλάχιστον ω το τέλο τη περίοδου των δημοσιονομικών προοπτικών, το 2013. Σα ευχαριστούμε για αυτέ τι διευκρινήσει, Επίτροπε. Κυρία Χούμπνερ. Δύο σύντομα θέματα. Ναι και κάθομαι δίπλα στον Πάτσι Λόπες. Θα ήθελα να πω ότι η χώρα των Βάσκων βρήκε ένα ιδιαίτερο τρόπο για να προχωρήσει. Και αυτή η ιδιαίτερη μεθοδολογία αποτέλεσε και την επιτυχία της χώρας των Βάσκων. Όταν πριν από μερικά χρόνια σκεφτόσαν το, το Μουσείο Guggenheim και αμφισβητούσαν πολύ το τι ρόλο θα παίξει στην ε, περιφερειακή ανάπτυξη. Αν σκεφτεί κανείς ε, την εικόνα που θα πρέπει να έχει μια περιφέρεια, ε, μπορεί να προσελκύσει όχι μόνο ο κόσμο για να την κατοικήσει στην περιοχή αυτή, αλλά και επενδυτές. Από την εμπειρία μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσα ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβαδίζει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ανάγκη να πείσουν τις περιφέρειες να γίνουν πιο ελκυστικές και να επενδύσουν στην αύξηση της, στη βελτίωση της εικόνας τους προκειμένου να προσελκύσουν κόσμο. Τώρα, το έλλειμμα ενημέρωσης είναι χρόνια νόσος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεκαετίες ολόκληρες το συζητούμε αυτό και μας προβληματίζει και ακόμη και σήμερα μας ταλανίζει το πρόβλημα της ελλειπής πληροφόρησης, ελλειπούς πληροφόρησης. Προσπαθούμε η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση να αναμειχθεί στη συζήτηση για την Ευρώπη και να μην μένθεται συνέχεια την Ευρώπη, αλλά να συμβάλλει στη, συνε... στη συζήτηση. Ο πολίτης όταν έχει προβλήματα θέλει να μπορεί να αποτανθεί σε κάποιον οικείο, σε κάποιον που μπορεί να εντοπίσει και να προσωποποιήσει και δεν θα πρέπει να ενδίδουμε στο παιχνίδι της ενοχής που είναι από τα αγαπημένα μας παιχνίδια, δηλαδή ο ένας να κατηγορεί τον άλλον ως ένοχο και να απεκδίεται των ευθυνών του. Σε ό,τι αφορά την επικουρικότητα. Η επικουρικότητα, όπως ξέρετε, είναι κάτι που εμπίπτει στις εθνικές αρμοδιότητες. Και υπάρχει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών λύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της επικουρικότητας. Τα τελευταία χρόνια όμως ε, υιοθετήσαμε μια στρατηγική προσέγγιση μιας ε, ισχυρής κεντρικής πολιτικής, αλλά μέσα σε αυτή την πολιτική πόλεις όπως η Δρέσδη και άλλες μπορούν να βρουν ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν και να εφαρμόσουν τη δική τους αναπτυξιακή στρατηγική, να εκπονήσουν προγράμματα, να διεκδικήσουν χρηματοδότηση γιατί καλή η διαρθρωτική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά θα πρέπει κάθε χώρα και κάθε βαθμίδα να βρει πώς θα την εφαρμόσει τοπικά. Ο πρόεδρος Βαντεμπράντε. Ο δήμαρχος της Μάλαγα έθεσε ένα σημαντικό ζήτημα. Όλοι θα θυμούνται το λόγο της Μάργαρετ Θάτσερ στην Πρίζ που έλεγε ότι οι αποφάσει για τη Μεγάλη Βρετανία πρέπει να λαμβάνονται στο Λονδίνο και ότι η επικουρικότητα φτάνει. Δεν θέλουμε άλλη. Τότε βέβαια γινόταν λόγος για εγκύτητα και επικουρικότητα. Οπότε, ναι, είμαι υπέρ της διαθεσμικής επαναξισορρόπησης και σε συνεργασία με τους τοπικούς δημάρχους. Ένα καλό παράδειγμα, ε, το η σύνοδος των δημάρχων για τις κλιματικές αλλαγές και τις ενεργειακές ανάγκες. Εκεί γίνονται προσπάθειες σε τοπικό επίπεδο, γιατί 70% των συνεπειών των κλιματικών αλλαγών γίνονται αισθητέ σε τοπικό ακριβώς επίπεδο. Έπειτα, κυρία Κρέλ, έχετε δίκιο. Πρέπει να ενημερώνουμε καλύτερα για το τι προέρχεται από πού. Και όχι απλώς να κάνουμε λόγο για το μεγάλο πρόβλημα επικοινωνίας. Υπάρχει πρόβλημα και το πρόβλημα είναι διορθωτικό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είναι, δεν είναι θεσμικά εφικτό να γίνει μια κοινή, ένα κοινό ανακοινωθέν ή ένα έγγραφο ενημερωτικό μαζί με το Συμβούλιο ή με την Επιτροπή. Διότι αυτό δεν συμφωνεί, δεν συνάδει με τους κανόνες. Θα πρέπει λοιπόν να καταστεί σαφές ότι υπάρχουν πράγματα προφανή και να ξέρουμε από πού προέρχονται τα μηνύματα. Χρησιμοποιούμε Μπορούμε μάλλον να χρησιμοποιήσουμε την εικόνα της Ένωσης, να την παρομοιάσουμε με ένα αυτοκίνητο. Πίσω βρίσκεται το Συμβούλιο, η μηχανή είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα καύσιμα είναι το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά για να λειτουργήσει ένα αυτοκίνητο και να τρέξει, να κυλήσει, χρειάζονται και ρόδες. Γι' αυτό έχουμε την Επιτροπή των Περιφερειών, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Δεν είναι λοιπόν μόνο μέρος του οχήματος οι περιφέρειες το κάνουν να τρέχει. Ας αλλάξει η μηχανή, ας αλλάξουν τα κάψιμα Αλλά οι ρόδες πρέπει να είναι εκεί. Και για την πρόθεση των νέων προϊόντων, για τα πιο ευέλικτα μέτσα και μέτρα. Ήθελα να θυμηθείτε τι είπε ο αντιπρόεδρος ε, σε μια τελευταία μας συνάντηση. Κάθε περιοχή, κάθε περιφέρεια έχει τουλάχιστον ένα πλεονέκτημα στα χέρια της. Πρέπει λοιπόν να τα ενώσουμε αυτά τα πλεονεκτήματα. Μόνο έτσι θα είμαστε βέβαιοι ότι θα βελτιώσουμε τα πράγματα, θα τα κάνουμε πιο καλά. Σας ευχαριστούμε, αλλά έχουμε περίπου κάνα δεκάλεπτο και έχω τουλάχιστον 5-6 ομιλητές που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα τους καλέσω λοιπόν να μιλήσουν και εάν μπορέσουν να είναι σύντομοι θα ακούσουμε και άλλους έναν-δυο. Ο Μέκλ Σνάιντερ λοιπόν, γραμματέας της Σαξονίας. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο εκ μέρους, της, ε, εκ μέρους του ΕΛΚ και της Επιτροπής ε, της Περιφερειακής Επιτροπής. Βεβαίως ε, θα πρέπει να έχουμε καλύτερη ενημέρωση στις προσεχείς εκλογές. Είναι κάτι που ήδη έχει λεχθεί. Ε, νομίζω ότι έχουμε διαλέξει πάρα πολύ καλά το θέμα μας, δηλαδή πρόκειται για μια παγκόσμια κρίση Πρόκειται για την παγκοσμιοποίηση και για τις περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια όμως έχει πληγεί σε διαφορετικό βαθμό και γι' αυτό χρειάζονται και διαφορετικές απαντήσεις. Γι' αυτό και θέλουμε να έχουν αρμοδιότητες οι περιφέρειες. Θα πρέπει να δικαιώσω την κυρία Χιούμπνερ. Έχουμε προοδεύσει πάρα πολύ κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, αλλά και πάλι θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία, να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στις περιφέρειες για να μπορέσουν πραγματικά να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την υπάρχουσα κρίση της παγκοσμιοποίησης. Επίσης ε, έχουμε θίξει το θέμα της κοινωνικής συνοχής και βεβαίως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Αν πάρουμε παραδείγματος χάρη μια περιοχή σαν δική μου ε, η οποία ε, υποφέρει από ορισμένε δομικές διαφροτικές αδυναμίες ε, και βεβαίως ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή με αυτούς οι οποίοι έχουν, είναι εξειδικευμένοι και με αυτούς οι οποίοι είναι ανειδίκευτοι. Οι ανειδίκευτοι απολύονται και εξειδικευμένοι δεν, δεν ξέρουν πού να δουλέψουν τελικά. Πρέπει να μεταναστεύσουν. Θα πρέπει να υπάρξουν νέε λύσει και μεγαλύτερη ευελιξία. Ο Λάμπερτ Βανίστελ Ευρωβουλευτής. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Βαντεμπράντεν αναφέρθηκε στον τομέα της καινοτομίας και βεβαίως είναι μια καινοτομία αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή εδώ. Συζητάμε μεταξύ μας σε αυτόν τον ναό της δημοκρατίας, σε αυτή την αίθουσα και βεβαίως πρόκειται για μια πραγματική καινοτομία, πρόκειται για μια νέα συζήτηση ε, που λαμβάνει χώρα εδώ. Είμαστε άνθρωποι, επικοινωνούμε μεταξύ μας ε, ο κύριος ε, Μπαρόζο είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειών. Όλοι θα πρέπει να, να δηλώσουμε μια μεγαλύτερη συμμετοχή. Δυστυχώς ε, δεν έχουμε μέχρι στιγμής τις απαραίτητες ε, απαντήσεις. Ε, θα πρέπει να συζητηθούν αυτά τα θέματα στις περιφέρειες. Οι περιφέρειες θα πρέπει να δώσουν την απάντησή τους στο θέμα της αλλαγής του κλίματος, στο θέμα της ανεργίας, στο θέμα της οικονομικής κρίσης. Και βεβαίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή ενέκρινε ένα προϋπολογισμό που αναφέρεται και σε αυτές τις δυνατότητες της συμμετοχής. Βεβαίω θα πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειών και θα θέλαμε να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι προτίθεται να κάνει, γιατί θα πρέπει να λάβουν μέρος όλες οι περιφέρειες. Σας ευχαριστώ. Η Κατρίν Γκρέσ... Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί μου δώσατε το λόγο. Θα ήθελα να αναφερθώ ε, στις ε, υπερπόντιες περιφέρειες αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επίσης και για την αναδιάρθρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των οποίο όπως λέγονται. Και αυτό γιατί υπάρχει μια μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης και αηφόρου ανάπτυξης. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξει και καινοτομία και αηφόρος ανάπτυξη, έτσι ώστε οι οικονομικοί πόροι, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα και, τους, και την οικονομία, να έχουν την απαραίτητη και σωστή συμμετοχή. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα πρέπει να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε το στόχο της ενεργειακής αυτονομίας θα πρέπει βεβαίως να λάβουμε υπόψη μας ε, το πόσο έχουν πληγεί αυτές οι περιοχές, οι περιφέρειες, οι υπερπόντιες περιφέρειες σε σχέση ε, με την αλλαγή του κλίματος. Θα πρέπει να προωθήσουμε τις δημοτικές, περιφερειακέ περιφερειακές αρχές. Θα πρέπει να δημιουργηθούν συνεταιρισμοί και θα πρέπει να υπάρξει μια κοινωνική, ε, μια κοινωνική ανάληψη των ευθυνών. Θα πρέπει να μπορέσουμε να αμφισβητήσουμε αυτά τα συστήματα που ισχύουν για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε νέα συστήματα. Θα πρέπει η οικονομική ανάπτυξη αυτών των περιφερειών να προωθήσει τα πλεονεκτήματα που έχουν αυτές οι περιοχές, πράγμα που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε αηφόρο ανάπτυξη και ανάκαμψη. Θα ήθελα λοιπόν να δω πώς μπορεί η περιφερειακή πολιτική να προωθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά μέσα στα πλαίσια της σημερινής συγκυρίας. Ένας ακόμη μιλήτης έχει μείνει στο κατάλογο. Α, Αρίστο Εβέλα, Ευρωβουλευτής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα δίκτυο μικρών τραπεζών στην Ευρώπη και υπάρχουν δυστυχώς όλο και πιο αυστηροί διεθνείς κανόνες ε, και θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη μας τις δυνατότητες που υπάρχουν ε, και θα πρέπει να συνταχθούν κάποιες εκθέσεις για αυτό το σκοπό. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, φροντίσει ώστε να μην είναι αυτοί οι κανόνες απαγορευτικοί για τη λειτουργία των μικρών τραπεζών γιατί οι μικρές αυτές τράπεζες παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να αντιμετωπιστεί η περιφερειακή κρίση. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Επιτροπή να λάβει υπόψη της, την ύπαρξη αυτού του προβλήματος των μικρών τραπεζών και τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν. Ε, θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει σε επαφή με τους εκπροσώπους αυτών των μικρών τραπεζών. Ακόμη κανένα δυο ερωτήσεις, αλλά πολύ σύντομες παρακαλώ. Ξέρω περιμένετε πολλή ώρα. Η κομμουνιστική ιδεολογία μου πίσω από την θέλησή μου να βλέπω καλοπροαίρετη, καλοπροαίρετο προβληματισμό για τα προβλήματα της κρίσης που έχουμε με σπρώχνει να βλέπω το κύριο τα τεράστια μέσα παραγωγής που υπάρχουν σήμερα σε όλη τη γη και διαρκώς εξελίσσονται και την κρίση πραγματικής υπερπαραγωγής που έχουμε που αυτά τα αγαθά που βγαίνουν δεν μπορούν να πάνε στους λαούς. Τελείως αντίθετο με την κοινή λογική να λύσει τα προβλήματα με τεράστιο κοινωνικό συντονισμό είναι το πλαίσιο σήμερα να λύνουν τα προβλήματα οι υπερεπενδυτές που κλέβουν και τα λεφτά όπως το είδαμε και σε αυτή την κρίση. Okay. Ε, ξέροντας, σας παρακαλώ, ξέροντας πως δεν συμφωνούμε, κάνω μία πρόταση. Σαν κριτήριο για τα μέτρα που παίρνετε, βάλτε δύο δείχτες ενδεικτικά τους λέω, ο ένας να είναι ποσοστό ε, όχι απασχολησιμότητας αλλά δουλειάς σε σχέση με τον ενεργό πληθυσμό και δεύτερο ποσοστό λαϊκής κατανάλωσης για τα 80 εκατοστά του πληθυσμού ποσοστό λαϊκής κατανάλωσης Δυστυχώς θα πρέπει να σας διακόψω που υπάρχει. Τέλειωσα. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε θερμά. Μία τελευταία πολύ σύντομη ερώτηση όμως, γιατί πολλά χέρια βλέπω, αλλά δεν θέλω να ευνοήσω μία πλευρά της ένωσης βάρος της άλλης. Μία τελευταία πολύ σημαντική ερώτηση και μετά θα ξαναδώσω το λόγο στα μέλη του πάνελ για τις τελικές απαντήσεις. Ευχαριστώ ε, κυρία Πρόεδρε για την δυνατότητα που μου να πάρω το λόγο. Είμαι δήμαρχος μιας μικρής πόλης ε, της Ιταλίας ε, μία από τις μικρές μικρές κοινότητες που υπάρχουν στην ε, Ιταλία. Άκουσα τις ερωτήσεις που τέθηκαν, άκουσα και τις απαντήσεις. Επιτρέψτε μου ε, να σας εκφράσω ορισμένες σκέψεις, ειδικότερα στον τομέα της έλλειψης της ενημέρωσης. Συγγνώμη, θα πρέπει να θέσετε μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση στο πάνελ αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι, ναι φτάνω, φτάνω και στην ερώτηση. Ε, σχετικά με την έλλειψη ενημέρωσης που υπάρχει ε, και που οφείλεται στην Επιτροπή. Είναι δυνατόν βεβαίως οι περιφέρειες παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Μπορούμε να αυξήσουμε τη συνειδητότητά μας και την ενημέρωση. Ε, αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να το πω στην Επιτροπή και επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα του πολιτισμού, στην κουλτούρα, στην πολιτιστική πολιτική που θα πρέπει να ασκήσουμε. Ε, Βεβαίω η κουλτούρα είναι, αποτελεί μια τεράστια πρόκληση και όλοι μας θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση. Λοιπόν, Ζητώ συγγνώμη αγαπητοί κυρίε και κύριοι που σας ζόρισα για να είστε πολύ σύντομοι αλλά ήθελα να μείνει λίγος χρόνος και στα μέλη του πάνελ για να απαντήσουν. Παρακαλώ ο κάθε πανελίστας να επιλέξει ποια απάντηση σε ποια ερώτηση θα απαντήσει. Ε, πολλή συζήτηση γίνεται για το κατά πόσο η κρίση θα αναδείξει μια ισχυρότερη, μια στενέστερη Ευρώπη. Η ισχυρότερη επειδή θα μπορέσει να συνεργαστεί ή πιο αδύναμη γιατί θα ενδώσει στον προστατευτισμό και θα υπονομεύσει την εσωτερική αγορά. Πώς θα μπορέσει η περιφερειακή πολιτική να συμβάλλει στο να εξέλθει ισχυρότερη από την κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι ασθενέστερη. 1,5 λεπτό μόνο στον καθένα έχει απομείνει για να απαντήσετε στις παρησίμαντες αυτές τις ερωτήσεις. Ο Επίτροπος Πάβελ Σαμέτσκι. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Σνάιντερ. Και επαναλαμβάνω αυτά που είπε. Χρειαζόμαστε περισσότερη ε, ελαστικότητα, περισσότερη απόδοση ευθυνών από την πλευρά των περιφερειών και μεγαλύτερη πειθαρχία. Σε ό,τι αφορά τι υπεραπόμακρε περιοχές, η πολιτική συνοχή λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ε, πολύ απομακρυσμένων περιοχών και να ενισχύσει τους δεσμού αυτών των περιοχών. Επενδύονται κονδύλια στο σκοπό αυτό. Είναι όντω δύσκολα τα προβλήματά τους, αλλά η πολιτική συνοχή τα συμπεριλαμβάνει και δεν τα παραμερίζει καθόλου. Τώρα, στο θέμα της Προέδρου. Δύο είναι τα επιτεύγματα της ε, πολιτικής συνοχής. Καταρχήν έμεσα υποστηρίζει τους εθνικούς προπολογισμού που αυτή τη στιγμή υφίστανται τεράστιες πιέσεις, οπότε δράβραχε πρόθεσμα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το δεύτερο επίτευγμα της πολιτικής συνοχής, μια και συμβάλλει στην υλοποίηση των βασικών στόχων των ε, σχεδίων οικονομικής ανάκαμψης. Επιμένει στη βελτίωση των υποδομών, στην ενίσχυση των ε, επενδύσεων και στην υποστήριξη του ανθρώπινου κεφαλαίου. Δίνει ευκαιρίες. Μπορεί να μην είναι αποφασιστικός παράγων, αλλά σίγουρα βοηθά η πολιτική συνοχής. Ευχαριστώ, Πρόεδρος Επιτροπής Περιφερειών φαντάζομαι δεν είναι έκπληξη το ότι συμφωνώ πλήρως και στενίζομαι απόλυτα αυτά που είπε ο Μάικλ Σνάιντερ. Θα πρέπει να υλοποιούμε με μεγαλύτερη ελαστικότητα τους στόχους μας ώστε να δίνουμε την σωστή απάντηση στην κατάλληλη στιγμή. Συμφωνώ και με τα σχόλια για τις κλιματικές αλλαγές. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Σε ό,τι αφορά τις... το δίκτυο των μικρών τραπεζών, σίγουρα είναι η εξουσία σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια της λειτουργίας τους, απόλυτη διαφάνεια και οι κανόνες να μην προσαρμόζονται μόνο στην ε, κάστοτε κατάσταση. Συνάδελφοι, ίσως θα πρέπει να υιοθετήσουμε και κάποια εναλλακτικά κριτήρια για την αξιολόγηση της κατάστασης. Και στη Γαλλία υπευλήθη πρόταση για την ε, υιοθέτηση νέων κριτήριων. Τέλος, στην ερώτηση του κυρίου Βανίστερ Ρόι, θα ήθελα να πω ότι η πρότασή σας ε, είναι πολύ καλή και θα μπορούσαμε να την ε, εφαρμόσουμε, να συνεργαστούμε εμπράκτως προκειμένου με εταιρική σχέση να εφαρμόσουμε μια λύση στις παγκόσμιες εκλογές. Επειδή η κυρία Τερίτο Χιούμπνερ θα λάβει το λόγο για να ολοκληρώσει μετά την ε, απογευματινή μας εναρκτήρια συνεδρίαση, θα δώσω πρώτο το λόγο στον πρόεδρο Πάτσι Λόπε. Δε και περισσότερες ερωτήσεις ε, αφορούσαν περισσότερο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρά εμάς. Θα ήθελα να συμμεριστώ κι εγώ μία πρόταση, μία διαπίστωση που ακούστηκε ότι η κρίση ως παγκόσμια χρήζει παγκόσμιων λύσεων. Αλλά χρειάζονται και τοπικές λύσεις, γιατί οι τοπικές λύσεις έχουν την δέουσα ελαστικότητα και μπορούν να προσαρμοστούν στην εκάστοτε πραγματικότητα ή στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να ληφθούν υπόψη οι τοπικές ανάγκες για να είναι αποτελεσματικές οι λύσεις. Γι' αυτό και είμαι υπέρ της ενίσχυσης της τοπικής εξουσίας των Δήμων, Κοινοτήτων και της Περιφέρειας θα πρέπει ταυτόχρονα να ενισχύσουμε και το τοπικό και περιφερειακό σκέλος, αλλά ταυτόχρονα να μην αμελήσουμε και το ευρωπαϊκό, γιατί αυτό μας δίνει την κάλυψη και δίνει τις βάσεις για μια αποτελεσματική απάντηση. Τώρα η Ντανίτα Χιούμπνερ, η κυρία Όρος μάλλον, πριν δώσουμε το λόγο στην κυρία Χιούμπνερ. Θα ήθελα να πω και εγώ ότι ε, ήταν ε, η απόφασή μας σαφής από όλες τις πλευρές. Ε, υπάρχει μια καταφατική απάντηση. Θέλουμε όλοι μας μια δυνατή Ευρώπη και βεβαίως η αλλαγή του κλίματος, η ενεργειακή κρίση, η οικονομική κρίση είναι προβλήματα τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όλοι. Υπάρχει ένα κοινό αίτημα σε σχέση με την κρίση που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να λάβουν μέρος όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των Δήμων, των κοινοτήτων, της περιφέρειας και βεβαίως μπορούμε μόνον όλοι μαζί και από κοινού να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Θα πρέπει να αναλυφθούν οι ευθύνε από όλες τις πλευρές. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι είμαστε εταίροι, ότι όλοι έχουμε κοινού στόχους, ότι έχουμε κοινέ υποχρεώσεις και έχουμε και την δυνατότητα μιας κοινή συμμετοχή. Και όλοι μαζί μπορούμε με τη συνεργασία μας να δώσουμε μια απάντηση. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ε, σαφές το μήνυμα και το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους ε, για τις ερωτήσεις σας, για τα σχόλιά σας ε, και βεβαίως πολλά θέματα θα συζητηθούν αυτές τις Open Days. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς οι οποίοι έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν και ιδιαίτερα όταν οι ομιλητές μιλούσαν πάρα πολύ ε, γρήγορα. Ε, θα δώσω το λόγο στην κυρία Χιούμπνερ η οποία θα κάνει ορισμένες τελικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ για αυτήν την ευκαιρία. Πάντοτε είναι καλό να μιλάει κανείς στο τέλος. Για όσους δεν πρόλαβαν, μην ξεχνάτε έχετε ακόμα τρεις μέρες για να λάβετε το λόγο. Θα έχετε λοιπόν ε, πολλές ευκαιρίες. Κάποια συμπεράσματα τώρα, κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με αυτά που πραγματικά είπατε όταν πήρατε το λόγο. Είναι σαφές ότι σήμερα δεν ξέρουμε ή τουλάχιστον δεν ξέρουμε αρκετά για τον αντίκτυπο της ε, σημερινής κρίσης σε περιφερειακό επίπεδο. Σίγουρα αυτό πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω και πρέπει να διεξαγάγουμε συμπεράσματα. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που η Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο θα κάνουν, αλλά και η Επιτροπή των Περιφερειών να καταλάβουν καλύτερα τους ερχόμενους μήνες ποια, ποιος είναι ο πραγματικός ε, αντίκτυπος της κρίσης στις περιφερειακές και τοπικές μας οικονομίες. Κάποιες περιοχές επηρεάζονται και πλήττονται περισσότερο από άλλε. Δεν ξέρουμε ακριβώ το συνολικό αντίκτυπο τη κρίση, εκτό μικροφόνο μελήτρια, στο επίπεδο θα ποικίλει σίγουρα με, ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό και θέλω να δώσω έμφαση εδώ είναι ότι σημειώνουμε το γεγονός ότι η κρίση έχει πλήξει τις τοπικές οικονομίες που ήδη είχαν πληγεί στο παρελθόν και έπειτα από τις διάφορους κλειδονισμούς λόγω των κλιματικών αλλαγών, των ενεργειακών προβλημάτων, των δημογραφικών πιέσεων. Καταλαβαίνω ότι ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων ε, πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού αν δεν θέλουμε να έχουμε ε, άλλους νέες αναταραχές εκ των υστέρων ως απόρρια της κρίσης. Ξέρετε καλύτερα κι εσείς τις περιφέρειες από ό,τι ξέρουμε εμείς εδώ στις Βρυξέλλες ότι το επίπεδο ε, των περιφερειών ε, ποικίλει ανά την Ευρώπη και δεν υπάρχει σαφής συσχετισμός μεταξύ του επίπεδου ανάπτυξης μιας περιφέρειας και της δυνατότητας απορρόφησης των ε, χτυπημάτων, των πληγμάτων από την κρίση. Θα πρέπει λοιπόν να το δεχτούμε ότι κάποιες περιφέρειες σίγουρα θα πληγούν περισσότερο, ίσως οι πιο κλειστές ή λιγότερο αναπτυγμένες. Θα δούμε πώς ε, τα καταφέρνουν οι περιφέρειες λοιπόν από μόνες τους, αλλά και τι μπορούν οι εθνικές πολιτικές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο να προσφέρουν αλλά να πω ότι και μετά την κρίση σίγουρα θα έχουμε ένα νέο χάρτη ε, περιφερειακό και τοπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να τον ε, μελετήσουμε προσεκτικά για να σχεδιάσουμε την επόμενη γενιά της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής. Όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στην Ευρώπη μετά την κρίση θα υπάρχει ακόμα το περιφερειακό και τοπικό στοιχείο πολύ ισχυρό. Κάτι άλλο που προκύπτει από τη σημερινή μας συζήτηση είναι ότι υπάρχει δυνατότητα σήμερα να ξανασκεφτούμε την πορεία που ασχοληθούμε για την ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό επίπεδο, αλλά και να αναθεωρήσουμε πολιτικές και εργαλεία ώστε να συνοδεύσουμε τις αλλαγές. Πάντως υπάρχουν πολλά διλήμματα. Υπάρχει το θέμα της εξέβρεσης της σωστής ισορροπίας μεταξύ των υφιστάμενων θέσεων εργασία λόγου χάρη και τη δημιουργία νέων, το πώ θα κινητοποιήσουμε τι εταιρείε και τι επιχειρήσει να επιβιώσουν από την κρίση, αλλά να τι προετοιμάσουμε να ε, κάνουν και την επιπλέον απόσταση που απαιτείται για να πάνε παραπέρα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια εδαφική προσέγγιση που να εντοπίζεται στο τοπικό στοιχείο και γι' αυτό είναι θετικό να ε, ζητούμε από τι κεντρικέ κυβερνήσει να σχεδιάζουν καλύτερα τη στόχευση των προτεραιοτήτων και όχι απλώς την διανομή των κεφαλαίων. Πώς θα συνδυάσουμε τις πολιτικές προτεραιότητες στο τοπικό επίπεδο, νομίζω ότι είναι καθοριστικό εδώ να καταλάβουμε τις τοπικές προτιμήσεις και να αξιοποιήσουμε την τοπική γνώση αλλά και όλα τα εργαλεία που έχουμε στο τοπικό επίπεδο. Και μια τελευταία κουβέντα επειδή όλοι ευχαριστούμε σήμερα την Ιρλανδία, να μην ξεχνάμε, μιλήσαμε πολύ για την επικουρικότητα, να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι η νέα περιφερειακή πολιτική παρατείνει και διευρύνει την αρχή της επικουρικότητας και στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Άρα και στι χώρε που υπάρχουν κυβερνήσει αλλά και όχι, θα υπάρχουν πολλέ δυνατότητε να εκμεταλλευτείτε αυτή τη νέα αρχή. Και αυτό το λέω για εσά που έρχεστε από τα πρώτα επίπεδα διακυβέρνηση και ζητάτε από εμά, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να συνεργαστούμε. Σα ευχαριστούμε λοιπόν ιδιαίτερω. Κλείνουμε την εναρκτήρια αυτή σύνοδο την, των Open Days, των ανοιχτών ημερών. Καταλήξαμε σε κάποια πρώτα συμπεράσματα και θα ήθελα να σα ζητήσω ευγενικά να αδειάσετε, να κενώσετε την αίθουσα, διότι το Ευρωκοινοβούλιο και η Επιτροπή του για την Περιφερειακή Ανάπτυξη θα συνεχίσει τις εργασίες της σε αυτήν την αίθουσα. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι και ελπίζω να σας ξανασυναντήσω τις ερχόμενες ημέρες. Ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε περαιτέρω στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης. Ευχαριστώ.